Good uh, Συνάδελφοι, καλησπέρα. Προχωρούμε στο σημείο 16 της ημερησίας διατάξεως. Προβλέπει η ημερησία διάταξη ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Σβάτσεμπερκ, Τον Εξωτερικών της Δημοκρατίας Τσεχίας για τις προτεραιότητες της Τσεχικής Προεδρίας. Να του ευχηθούμε ε, ένα θερμό καλωσόρισε Έχετε ξανάρθει βέβαια, αλλά όχι ως προεδρεύων του Συμβουλίου. Ε, για μας είναι μεγάλη χαρά να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Έχουμε και μια σχετική αντιπροσωπεία ε, και στο πλαίσιο των εργασιών της οποίας επισκεφθήκαμε την Πράγα όπου και σας ε, συναντήσαμε. Επίσης πρέπει τον ε, Υφυπουργό τον κύριο Γιάννη Κόχουτ να τον καλωσορίσουμε. Είναι ο υφυπουργό η ΙΦΙΠΕΞ. Και ε, πρέπει να υποδεχθούμε και να ευχηθούμε καλωσόρισαν κάποιους γερουσιαστές. Πέλοβα, Γίζνεκ και Γκρούτιχ. Καλωσορίσατε και οι τρεις. Κύριε Υπουργέ. γνωρίζουμε ότι έχετε τάξει ένα πρόγραμμα φιλόδοξο για την Προεδρία σας. Πολλές φορές βέβαια η ζωή και οι εξελίξεις ζωντανές ξεπερνάνε τις φιλοδοξίες μας στο πρόγραμμά μας. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η συγκυρία. Οι προτεραιότητές σας για την Επιτροπή μας είναι σημαντικές γιατί αφορούν την ε, εταιρική σχέση προς Ανατολάς, την ε, υπερατλαντική συνεργασία, ενεργειακή ασφάλεια. Για ε, αναφέρω μόνο τα θέματα εξωτερική πολιτικής του προγραμματός σας τις δύο τελευταίες εβδομάδες είδαμε κάποιες εξελίξεις που έλαβαν χώρα όσον αφορά την ανατολική την προσανατολάς πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης γίναμε μάρτυρες κάποιων ε, πάρα πολύ συγκλονιστικών εξελίξεων και συναισθηματικά φορτισμένων όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια. Είδαμε την επίσκεψη της Τρόικας ε, στην Λωρίδα της ε, Γάζης και αυτό το θέμα είναι θέμα το οποίο καίει την Επιτροπή μας. Είχαμε όμως αυτή την προστριβή για το αέριο, είχαμε και τι εξελίξει στην Γάζα, πολύ ενισχυτικά σοβαρά θέματα και σας ευχόμαστε καλό ταξίδι στα ταραγμένα νερά της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης κατά αυτή την, καθό το εξαήμερο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε και να ενημερωνόμαστε, να σας ενημερώσουμε πίσω όπως πάντα γίνεται Ήδη τα είπαμε πάρα πολύ καλά κατά την ε, επίσκεψή μας τότε στην Πράγα όπως προείπα. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που με καλέσατε σε αυτή την επιτροπή σας. Είναι πολύ σημαντική επιτροπή. After the ratifying of the Νομίζω ότι θα έχετε ακόμη πιο σοβαρέ αρμοδιότητε μετά την επικύρωση τη ε, συνθήκη τη Λισαβόνα. Επίση, θέλω να σα πω ότι κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό για οποιαδήποτε κυβέρνηση ε, είναι αυτό το πώς θα πάει η θητεία της στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση αυτή η δημιουργική αντιπαράθεση με το Κοινοβούλιο με τις σκληρές δύσκολες ερωτήσεις γιατί έτσι κανείς προσγιώνεται από τον υψηλό πολλές φορές κόσμο των υπηρετικών υποθέσεων στην σκληρή πραγματικότητα. Έχουμε εδώ μια ολόκληρη πλημμυρίδα γεγονότων, μια χιονοστιβάδα γεγονότων που μας ε, υποδέχθηκαν με την αρχή του 2009 απαιτούνται ταχείες λύσεις θα πρέπει να πετύχουμε αποτελέσματα όσο γίνεται πιο γρήγορα βεβαίως εμείς ε, ακόμα είμαστε νέο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οπότε για μας αυτό είναι μια τεράστια υπόθεση Πάντως εμείς είμαστε βέβαιοι θα ανταποκριθούμε εις τις προκλήσεις που μας περιμένουν. Για την Γάζα. Είναι προτεραιότητά μας να υπάρξει κάποια λύση. Έστω και προπόθεσμα Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να άρουμε αυτή την ε, ανθρωπιστική τραγωδία και καταστροφή και να υπάρξει μια εξέλιξη, μια διαδικασία πολιτική πάρα πολύ βέβαια ε, ε, περίπλοκα είναι τα πράγματα έχουμε το Ιράν το οποίο επηρεάζει τις εξελίξεις έχουμε τη Χαμάς και εμείς με τη σειρά μας θα πρέπει να δούμε τον πρόεδρο Αμπάς την Αλφατά με την νόμιμη κυβέρνηση της Παλαιστινικής Αρχής να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για μας ε, η δυτή, η, η δύο επιπέδων λύση είναι πιο σωστή. Έτσι πιστεύουμε θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει τους, ε, τις δύο πλευρές να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι να συμμετήσουν. Θα πρέπει επομένως να υπάρξει μια πρακτική απτή διαδικασία ή προσέγγισης ε, της Αραβικής Ένωσης αμέσως τη βοήθεια θα πρέπει να έχουν και τη Αιγύπτου. Βεβαίως. Δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι η λύση πάντοτε θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους εμπλεκομένους. Βεβαίως και προϋπόθεση απαραίτητη είναι η εκεχηρία, η πάυση του πυρός. θα πρέπει να αποσύρει να του το Ισραήλ και τη Χαμάς επίσης να πάυσει τις αυτοπαξίες την πλευρά της. Η Τρόγιο αμέσως μόλις άρχισαν τα γεγονότα επισκεφθήκε την πλευρά της Γάζας, φρόντισε για να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια και συνέβαλε στο να υπάρξει τρίωρη και πρόβλημα σε δύο ανακοινώσει και ετοιμάσαμε μία μέση διάταξη για το Συμβούλιο. Επιβάλλεται να ασχοληθεί το Συμβούλιο που είναι σήμερα η κατάσταση και να υπάρξει κάποια προοπτική για βαθμία επίτευξη της επιτυχίας. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την εμπλοκή του Προέδρου Αμπάς αλλά και να καταλήξουμε σε ένα βιώσιμο πολιτικό κράτο, το οποίο να μπορεί να ζήσει με ειρήνη και ασφάλεια πλάι πλάι με του Ισραηλινού. Είπαμε να υπάρξουν τρει παρατηρητέ από το τσεχικό ΙΤΑΞ. Αυτό συμφωνήθηκε και ήδη αυτοί έχουν αναχωρήσει για να μεταβούν Βεβαίως και θα είναι σε επαφή με όλες τις μη οργανώσεις, με τους διεθνείς φορείς, με την Επιτροπή του Ερυθροσταυρού και όλους γενικά. Και έτσι και θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να φροντίσουμε αυτά τα οποία άμεσα τώρα χρειάζονται. Τι θέλουμε να πετύχουμε τελικά, να υπάρχει ένας εύρεθμος έλεγχος διεθνής της καταστάσεως κυρίως όσον αφορά τη Γάζα, τη Γάζα γιατί αυτό πρέπει να υπάρχει παραγωγή των συνόρων γι' αυτό θα πρέπει να είναι δυνατόν κανεί να μπορεί να χρησιμοποιήσει και την θάλασσα ε, όσον αφορά την αποθάλασσα προσέγγιση όσον αφορά τους Ισραηλινού, θα πρέπει να ανοίξουν τα συνοριακά περάσματα θα πρέπει να αρθεί ε, το, το, το σημερινό εμπάργο ήδη εμεί έχουμε προσπαθήσει να πείσουμε το Ισραήλ να ανοίξουν τα περάσματα να είναι έτοιμο το Ισραήλ να αναπτύξει ε, ό,τι χρειάζεται για να μπορέσουμε να έχουμε φυσιολογική φυσιολογικό ανοίγμα των συνόρων θέλουμε να υπάρξει βαθμία συμφιλίωση με τους Παλαιστινίους οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί όσον αφορά την Χαμάς και τους ε, καταβλισμούς, οικισμούς των Παλαιστινίων. Άλλη μια πρόκληση βεβαίω και είναι η ενεργειακή ασφάλεια και σας υπενθυμίζω ότι η τσεχική προεδρία και πριν αλλά το μάλλον τώρα επιμένει ότι κατεπηγόντως Χρειάζεται μια κοινή πολιτική για την ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κόστος του να μιλήσουμε αυτή την πρωτοβουλία θα είναι πάρα πολύ ψηλό. Για μας αυτό είναι η προτεραιότητα. υπάρχει εναλλακτική προμήθεια του φυσικού αερίου, δηλαδή τι έγινε με την Ουκρανία, δηλαδή τι έγινε με τις τιμές, οπότε το πολλά κάνει όσο πιο με τις ενέργειες μπορεί. Είδατε τώρα πρόσφατα ε, ότι αυτά τα οποία έγιναν τώρα έχουν ξεπεραστεί και ήδη το αέριο έχει φτάσει σε ελεύθερη παροχή στην Σλοβακική Μεθόριο. Ρωσία και Ουκρανία δεν είναι αξιόπιστοι προμηθευτέ. Αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούμε για να βρούμε εναλλακτικού προμηθευτέ και εναλλακτικού αγωγού. Άρα το Ναμπούκο είναι κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά την κυριότητα των έργων υποδομής στην Ευρώπη γιατί θα πρέπει να αρθεί ο κίνδυνος που υπάρχει όσον αφορά το ότι κάποιες τρίτες χώρες ε, έχουν δυσκολία προσβασιμότητα στην αγορά και γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ε, δεν θα πέσουμε στα νύχια κάποιων ε, εταιριών ή κάποιων που γενικά θα εξυπηρετούν τα πολιτικά του συμφέροντα. Θα πρέπει επομένω να συνεχίσουμε να διευρύνουμε, να βαθύνουμε τη συζήτηση για το ενεργειακό. Άρα να συνεχιστεί ο διάλογος με τη Ρωσία γιατί αυτό είναι προ το συμφέρον όλων της Ρωσίας συμμενοβαλλομένες. Να υπάρχουν επαφές έντονες και δημιουργικές Όμω σε μια νέα φάση εταιρική σχέση και συνεργασία με τη Ρωσία. Βασικό στόχος της Προεδρία είναι η πολιτική ηγετνίασης και εταιρική σχέση με την Ανατολή. Να αναβαθμιστεί η συνεργασία με την Ανατολική Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε. Μια τέτοια συνεχτική πολιτική με τις σχετικές χώρες. Αυτό δεν θα καθορίσει μόνο την ποιότητα των σχεσιών μας, αλλά θα βελτιώσει και το βιωτικό επίπεδο των χωρών. Γι' αυτό και θα πρέπει να δούμε το θέμα ε, πιο αναλυτικά στα τέσσερα εξή κεφάλαια ότι αυτή η εταιρική σχέση δεν αποτελεί απειλή για κανένα. Είναι μια θετική επικοδομητική πολιτική των 27 κρατών μελών προς τις έξι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Είναι, όπως έχουν σήμερα οι δημοσιονομικές προοπτικές, είναι ουδέτερη πολιτική όσον αυτόν τον προπολογισμό. Δεν χρειάζονται τίποτε κεφάλαια τα οποία θα πρέπει να εκταμιευτούν, τα οποία θα πρέπει να δεσμευτούν στον προπολογισμό για να προχωρήσει αυτή η συνεργασία. Άρα το κόστος ε, είναι αμεληταίο σε σχέση με το κέρδος, την ωφέλεια που θα αποδώσει αυτή η εταιρική σχέση. Με τίποτα επίσης αυτή η πολιτική δεν πρόκειται να γίνεται εις βάρος ε, εταιρικής σχέση με άλλες χώρες. Θα συμπληρώσει ε, τις περιφερειακές υπάρχουσες πολιτικές. Ούτε αποτελεί ένα φτηνό εγκαταστατό της διεύρυνσης. Είναι κάτι το οποίο γίνεται ε, κατά παραγγελία ο Ρωσιπίν για την περιοχή αυτή που, που το χρειάζεται για να τους φέρει ευημερία και σταθερότητα. Υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό θέμα που πρέπει παρακάτω να μας απασχολήσει. Είναι η Ευρώπη και σχέσεις με τα Δυτικά Βαλκάνια. Μια που η πρόοδος, η σύνδεση, η προσέγγιση των Δυτικών Βαλκανίων με την Ένωση είναι μια προτεραιότητα κλειδί για την Προεδρία μας. Πάντα για την εξωτερική μας πολιτική. Είναι θέμα κατεπήγων όπως και άλλα τα οποία θα πρέπει παραλύρου να τα φροντίζουμε. Ε, τα Βαλκανία έχουν, το ξανατονίζουμε, ευρωπαϊκή προοπτική και η Προεδρία μας προτίθεται να σημειώσει πρόοδο στο θέμα τούτο. Να πλησιάσουν περισσότερο οι χώρες αυτές στην Ευρώπη. να αναβαθμιστεί το καθεστώς των υποψηφίων. Μετά το Μαυροβούνιο, το οποίο υπέβαλε τη θέση του για να ενταχθεί στην κοινωνία το, το Δεκέμβριο του 2008, έχουμε και άλλες χώρες οι οποίες ακολουθούν και θα κινηθούν τον τρόπο κατά την Προεδρία μας. Εμείς καταβάλουμε πάσα προσπάθεια για να δοθεί συνέχεια σε αυτή την αίτηση με τις δέουσες διαδικασίες και οι εμπειρογνώμονε τη Κομισιόν θα πρόκειται να αξιολογήσουν το επίπεδο ετοιμότητο αυτών των χωρών. Επίση θα ζυγίσουν και θα αποτιμήσουν τι μεταρρυθμίσει που έχουν προβεί αυτέ οι χώρε επίση. θέλουμε να συνεχιστεί η βοήθεια με στόχο την σταθεροποίηση κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των χωρών αυτών και στο Πεσυφοπέδιο επίση, ε, έχουμε και την αποστολή Ρελέξ θεωρούμε ότι είναι το μήμα των Δυτικών Βαλκανίων το Πεσυφοπέδιο και συνεχίζει να αξίζει την αμέσως προσοχή της Ένωσης. Η Κομισιόν ανέλαβε και εξεπώνησε μελέτη στον σύμφωνο σταθερότητας και σύνδεσης σε σχέση με τη χώρα εκείνη. Βεβαίω και το ότι υπάρχει οικονομική κρίση στην Ευρώπη αυτό επηρεάζει και το κοσμοπέδιο και τις ε, γειτονιάζουσες χώρες. Η Δυτική Ευρώπη τώρα που έχει κρίση χτυπάει το οικονομικό σοφοπέδιο που εξαρτάται τόσο πολύ και ήδη έχουν εκεί 60% ανεργία και άρα η χώρα αυτή θα έχει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στο μέλλον. διατλαντικές σχέσεις. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η ΕΠΑ είναι εταίροι πάρα πολύ σημαντικοί στον κόσμο. Γενικά κανένα σήμα και ευθυγραμμίζονται, αλλά υπάρχουν και κάποιε διαφοροποιήσει βέβαια. Οπότε η Συνδική Προεδρία θέλει να εδραιώσει αγαστέ σχέσει μεταξύ ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και Τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ γιατί θα πρέπει να επιβεβαιωθεί το πόσο σημαντική ε, ε, είναι η εταιρική σχέση των ΗΠΑ. Αυτό θα είναι το μήμα του έργου που πρέπει να επιτελέσουμε. Και γι' αυτό και του ζωμούντρου του θα αρχίσουμε επαφές αρχές Φεβρουαρίου πρόκειται να μεταβούμε ή στην ε, Washington τόσο ώστε να παρουσιάσουμε αυτές τις προτάσεις στη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ και η πρόθεσή μας είναι να συναντήσουμε κόσμο από το Υπουργείο Εξωτερικών, από την Βουλή των Αντιπροσώπων, από τη Γερουσία και στα πλαίσια της Προεδρίας επίσης θα οργανώσουμε επίσκεψη του Μπαράκ ή στην Ευρώπη. Άλλωστε θεωρώντας είχε εξηγωστεί παιδιά του ΝΑΤΟ. Για μην πούμε για την κλασική συνάντηση ε, ΝΑΤΟ, είπα, στο κατάλληλο της ε, Προεδρίας μας. Γιατί το Υπερταντικό Συμβούλιο είναι νέος μηχανισμός συνεργασίας. Αυτό έχει πια εδραιωθεί. Οπότε για αυτό και θέλουμε να μείνει ζωντανό το ενδιαφέρον του νέου Προέδρου για όλες τις δραστηριότητε μας. Βεβαίω και θα ασχοληθεί το Συμβούλιο, επομένω, με αυτά τα ζητήματα, με την εταιρική συνεργασία, την υπερατλαντική, γιατί βέβαια εδώ δεν έχουμε μόνο τη ΣΥΠΑ. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει και ο Καναδά, γιατί με τη χώρα αυτή έχουμε πάρα πολλέ κοινέ αξίε και κοινά πολλά οικονομικά συμφέροντα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας και τώρα θα περάσουμε στο συνηθισμένο γύρο ερωτήσεων από τα μέλη. Επειδή υπάρχουν πολλοί που επιθυμούν να ρωτήσουν, να περιορίσουμε το χρόνο ομιλίας σε 1,5 λεπτό. Ο κύριος Αλαφράνκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κύριε Υπουργέ να σας καλωσορίσω εξ ονόματος του ΕΛΚ και θα ήθελα να σε ευχηθώ καλή επιτυχία για την θητεία σας. Θα ήθελα να πω ότι μας άρεσε η πρόθεσή σας να επικυρώσετε το ταχύτερο δυνατό τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και θα ήθελα τώρα στο πλαίσιο αυτό να διατυπώσω ορισμένες ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά την κατάσταση της Γάζας και είναι αλήθεια ότι τα συμβάντα με τον μεγάλη ταχύτητα Κύριε Υπουργέ, υπάρχει δυνατότητα, όπως εκφράστηκε από διάφορους πρωθυπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αρθεί το εμπάργκο στη Γάζα, σε... ούτως ώστε να υπάρξει μια προσωρινή κυβέρνηση και υπάρχει και η δυνατότητα να αποκλειστεί, να αφαιρεθεί η Χαμάς από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων της Ευρώπης υπό την προϋπόθεση ότι ε, δεσμευθεί να, να σταματήσει τις τρομοκρατικές ε, πράξεις και να δεχθεί τη δημιουργία ενός Ισραηλινού κράτους. Ο Γενικός ε, Γραμματέας των Διεθνών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας μίλησε για την Ένωση για την Ανατολή και εξέφρασε τη δική του επιθυμία να υπάρχει ταχεία εξέλιξη πριν από το τέλος της θητείας της παρούσας Κομισιόν σε μια, συμφωνική, σε μια συμφωνία. Είναι η Τσεχική Προεδρία διατεθειμένη να κινητοποιήσει όλα τα μέσα υπέρ αυτής της προτεραιότητας και θα ήθελα να θίξω τώρα τις σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Η Χίλαρη Κλίντον είπε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν θα μπορέσουν από μόνε του να επιλύσουν όλα τα προβλήματα τα οποία θέτει ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Αλλά και ο κόσμο δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα αυτά χωρί τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορούσατε, κύριε Υπουργέ, πέρα από τι συναντήσει που έχουν προβλεφθεί και από τι καλέ ε, προθέσει να βελτιωθούν αυτέ οι σχέσει, να μα προτείνετε κάποιο κατάλογο συγκεκριμένων ε, ε, δράσεων σε σχέση με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σαλαφράνκα. Κυρία Ντεκάιζερ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα εξ ονόματο τη ομάδα να σα καλωσορίσω και όπω ο κύριο Σαλαφράνκα θα ήθελα να πω ότι η προεδρία σα πραγματικά θα είναι πιο ευίωνη. Θα ήθελα να θέσω πρώτη, η πρώτη μου ερώτηση ήταν αυτή ακριβώς που έθεσε ο κύριος Σαλαφράγκα όσον ε, αφορά την άρση του εμπάργκο. Οι δύο άλλες ερωτήσεις ε, έχουν ως εξής. Η πρώτη αφορά την παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου που αναφέρει ο Επίτροπος κύριος, παρέφερε ο Επίτροπος κύριος Μισελ και οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί. Τι προτίθεται να κάνει η Τσεχική Προεδρία όσον αφορά αυτές τις καταγγελίες των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου και ποιες ποιες θα είναι οι επιπτώσεις όσον αφορά τις συμφωνίες σύνδεσης. Δεύτερον, υπήρχαν τρομακτικές καταστροφές ε, στη Γάζα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να υπάρξει μια εξεταστική επιτροπή η οποία να καταρτήσει έναν πλήρη κατάλογο. Το ερώτημα που θέτουν οι πολίτες της Ευρώπης είναι κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανεκοδομήσει τα όσα έχουν καταστραφεί χωρίς να ζητήσει το λογαριασμό από το Ισραήλ. Ε, τι θα γίνει, ποιο θα πληρώσει για την αποκατάσταση όλων αυτών των ζημιών, θα είναι το Ισραήλ ή όχι. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κάιζερ, ο κύριος Κάτσινγκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ και εγώ εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας θα ήθελα να σε ευχηθώ καλή επιτυχία στην επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας την οποία πραγματικά χρειαζόμαστε απαραίτητος Ιδιαίτερο σε αυτές τις εποχές της πολιτικής και οικονομικής κρίσης. Θα ήθελα να σας υποβάλω δύο ερωτήσεις και οι δύο αφορούν τα Δυτικά Βαλκάνια. Δηλαδή, τι προτίθεται να κάνει η Τσεχική Προεδρία για να βοηθήσει την Κροατία ούτως ώστε να διευθετήσει τα προβλήματα με τους γείτονές της προσβοράν γιατί με τον τρόπο αυτό η, συνέχιση των διαπραγματεύσεων δεν, ήταν εφικτή, δεν είναι πλέον εφικτή. Και οι δύο υποψήφιες χώρες θέλουν να προσφύγουν η μία κατά της άλλης στο δικαστήριο της Χάγης λόγω των εγκλημάτων από τον τελευταίο πόλεμο. Ε, τι θέλετε να πράξετε πώς θα λένε γεννηθείτε σε αυτή την περιοχή, ούτως ώστε να δώσετε αυτή, τη δυνατότητα σε αυτές τις δύο χώρες να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. E, θα ήθελα κατ' εξαίρεση ε, να σας ε, καλωσορίσω θερμά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ μέρους της ΟΕΝ. Όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική, κάθε φορά που υπάρχει κάποια κρίση, ε, γίνονται πολλές ε, δηλώσεις ε, για τον αγωγό Ναμπούκο αλλά και για την πολιτική που χαράστηκε γενικότερα. Η κρίση μοιάζει να βαδίζει προς το τέλος της. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν οι απαραίτητοι μηχανισμοί <clears throat> για να απευθυνθούν τέτοιου είδου καταστάσει στο μέλλον. Και θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσον προτίθεστε να αναλάβετε μακροπρόθεσμε πρωτοβουλίε που θα μα βοηθήσουν να αποφύγουμε παρεμφερεί καταστάσει στο μέλλον. Κυρίω ε, βήματα προ την κατασκευή επιτέλου του Ναμπούκου και ε, προ την ύπαρξη ε, πραγματικά μια σωστή ενεργειακή πολιτική. Ο κύριο Χωράτσεκ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό και την Προεδρία της Τσεχίας εκ μέρους της πολιτικής μας ομάδας. Ε, ακούσαμε ότι δολοφονήθηκε η συνεργάτης ε, στη Ρωσία, η συνεργάτης του γνωστού ε, ειδησιογραφικού πρακτορείου και της Άννα Σύμφωνα λοιπόν με τις ε, συμφωνίες που υπάρχουν στη Συμβουλή της Ευρώπης, η Ρωσία πρέπει να αναλάβει μέτρα έτσι ώστε να προστατεύσει τους ανθρώπους και να στηρίξει την εργασία τους. Η δική μου λοιπόν η ερώτηση είναι προς την Τσεχία όσον αφορά στις σχέσεις με τη Ρωσία και ρωτώ τι προτίθεστε να κάνετε έχοντας κατά νου ε, τα τελευταία γεγονότα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη στον τομέα της ενέργειας. Πληροφορίες φέρουν τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας, τον κύριο Νευτογάν, να έχει κατά τις χθεσινές του επαφές στις Βρυξέλλες απειλήσει ότι θα παρεμβάλλει εμπόδια στην κατασκευή του αγωγού του Ναμπούκο σε περίπτωση που στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανοίξει το κεφάλαιο για την ενέργεια. Όπως είναι γνωστό, ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κυπριακή Δημοκρατία, ενίσταται στο άνοιγμα του κεφαλαίου αυτού. Και αυτό γιατί κατά τις πρόσφατες έρευνες που διενήργησε η Κύπρος για εξέβρεση κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην οικονομική της ζώνη, η Τουρκία την απείλησε με τη λήψη στρατιωτικών μέτρων. Η ερώτηση μου είναι πώς προτίθεται η Προεδρία σας εν ώψη αυτών των δεδομένων να αντιμετωπίσει τις απειλές του κυρίου Ερτογάν για τον Αμπούκο Pipeline, line, και δεύτερο την απέτηση του για άνοιγμα του κεφαλαίου για την ενέργεια. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά το Παλαιστινιακό. Εν ώψη των παραβιάσεων του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου από τις Ισραηλινές αρχές στα Παλαιστινιακά εδάφη, με τον αποκλεισμό των κατοίκων της Γάζας, με την αύξηση του επικισμού στη Δυτική Όχθη, με την κατασκευή τείχου στα Παλαιστινιακά εδάφη για τον έλεγχο της περιοχής από τις Ισραηλινές αρχές, με τη σύλληψη και φυλάκιση πέραν των 10.000 Παλαιστινίων, με τους περιορισμούς που θέτει στην ελεύθερη διακίνηση των πολιτών, και εν ώψη της πρόσφατης επίθεσης στη Γάζα, που αποτέλεσε την πιο αιματηρή επιχείρηση των Ισραηλινών αρχών στα Παλαιστινικά εδάφη, πώς προτίθεστε να, να πράξετε σχετικά με την υπάρχουσα Συμφωνία Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ, καθώς και με τη διαδικασία αναβάθμισης των σχέσεων με το Ισραήλ. Ευχαριστώ. Thank you. This was the first... Αυτός λοιπόν ήταν ο πρώτος γύρος των ερωτήσεων. Κατά το δεύτερο γύρο θα είμαι πιο αυστηρός, θα περιορίσω το χρόνο σας σε 1,5 μόνο λεπτό. Ε, τώρα λοιπόν ο κύριος Υπουργός ε, θα απαντήσει ερωτήσεις. Όσον αφορά την κυβέρνηση, την προσωρινή κυβέρνηση ε, στην Παλαιστίνη, υπάρχει νόμιμη κυβέρνηση του κυρίου Αμπάς που την έχει αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται με προσωρινή κυβέρνηση, λέει ο μιλητής. Όσον αφορά τη Χαμάς, αν η Χαμάς αποκηρύξει την τρομοκρατία και δεχθεί τις γενικότερες ισχύουσες αρχές, τότε μπορεί να ξεκινήσει η πολιτική συζήτηση. δεν θα ήταν το πρώτο παράδειγμα ε, τρομοκρατικού κινήματος. Έχουμε προηγούμενο και στην Ιρλανδία. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι ε, υπάρχει εξέλιξη και αν τελικά η Χαμάς κατορθώσει να εξελιχθεί σε πραγματικό πολιτικό κίνημα δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Όμως για να γίνει αυτό πρέπει να αποκηρύξει η Χαμάς την τρομοκρατία. Δεν ξέρω τώρα ότι ε, μπορώ να τοποθετηθώ στην ε, συμφιλίωση των ίδιων των Παλαιστινίων μέσα στο, στο, στους κόλπους Παλαιστινίων. Όλοι το ευχόμεθα. Αυτή τη στιγμή τον σημαντικότερο ρόλο τον παίζει η Αίγυπτος, η οποία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, τότε ακριβώς κατέρευσαν οι συζητήσεις ανάμεσα στην Αλφατάχ και τη Χαμάς. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει, αλλά κατ' ουσίαν εδώ πρόκειται για ένα ενδοπαλαιστινιακό πρόβλημα. Όπως λοιπόν ε, ήδη ανέφερα κατά την ομιλία μου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αίτημα για αύξηση των κονδυλίων που θα μπορούσαν να επενδυθούν στην ε, ανατολική εταιρική σχέση. Για να είμαστε σαφείς, αυτήν την ε, πρωτοβουλία, ε, αυτή η πρωτοβουλία δεν θεωρούμε ότι πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία νέων θεσμών, κάτι το οποίο πάντα απαιτεί ε, αύξηση κονδυλίων. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι υπάρχουν προγράμματα. Ήδη υπάρχουν αρκετά προγράμματα και θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερο συντονισμό αυτών. Αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει ανάγκη εκταμείευση μεγαλύτερου αριθμού κονδυλίων. Όσον αφορά τις σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε. όπως σας είπα, τον επόμενο μήνα θα πάω στην Ουάσιγκτον Πιστεύουμε ότι όταν ο κύριος Ομπάμα ε, θα έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα θελήσει να επισκεφθεί στην Ευρώπη με θα θελήσει να επισκεφθεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ε, στο πρόγραμμα και η συνάντηση κορυφής με τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου ε, θα συζητηθούν κεφαλαιόδους σημασίας θέματα όπως είναι η κατάσταση στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν βέβαια. Πρέπει να συζητήσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες τη ε, διαδικασία ειρήνευσης ε, στη Μέση Ανατολή γιατί οι τελευταίες εβδομάδες κατέδειξαν ότι το θέμα αυτό έχει λάβει επίγουσα μορφή. Βεβαίως πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα με το Ιράν και με την ανάπτυξη πυρηνικών σταθμών. Άρα δηλαδή αυτά είναι τα σημαντικότερα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Θα ήθελα να απευθυνθώ στην κυρία Ντεκάιζερ. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Προεδρία δεν πρέπει να λειτουργεί ως δικαστής. Εγώ δεν είδα να έχει υπάρξει ποτέ πόλεμος όπου να γίνεται απόλυτα ε, σεβαστά, να γίνονται απόλυτα σεβαστά τα ανθρωπιστικά δικαιώματα πράγματι είναι απαραίτητο στη Γάζα ε, να δοθεί άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια και μετά να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση της περιοχής. Εάν πράγματι διαπιστωθεί ότι υπήρξε παραβίαση ε, του ανθρωπιστικού δικαίου, τότε ε, θα πρέπει να δούμε ε, τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά πρώτα πρέπει να επιβεβαιωθούν αυτές οι υποψίες και μετά θα συζητήσουμε για τον δεχόμενο των κυρώσεων. Πρόκειται να συζητήσουμε πρώτα με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών ε, θα συζητήσουμε την άλλη, το άλλο βράδυ με τον Άραβα Υπουργό Εξωτερικών σε δύο διαφορετικές τελείως συναντήσεις και βραδιές. Αυτό θα γίνει στις Βρυξέλλες. Πάντως, ε, οτιδήποτε μπορεί να γίνει στη Γάζα, οποιασδήποτε σε ανθρωπιστική βοήθεια, Προς το παρόν τουλάχιστον χρειαζόμαστε υποστήριξη και ε, χρειαζόμαστε και κάποια ε, καλή βούληση εκ μέρους του Ισραήλ. Πρέπει λοιπόν να έχουμε στενές επαφές και με το Ισραήλ και με τα αραβικά κράτη. Αυτά τα προβλήματα δεν είναι τα πιο εύκολα θα έλεγα, αλλά είμαστε σωστά προετοιμασμένοι. Ε, ως τον κύριο Κατσίν. Κατά την ε, παρουσίασή μου σας είπα αναφέρθηκα στα προβλήματα των Δυτικών Βαλκανίων. Στόχος μας είναι όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να τις φέρουμε όσο πιο κοντά γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τελικό στόχο κάποια στιγμή όλα αυτά τα κράτη να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού. Αυτή τη στιγμή η Κροατία είναι η καλύτερα προετοιμασμένη χώρα και αναμένουμε όλοι μας να συνεχιστεί ε, με ήπια μορφή η διαδικασία ένταξής της. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι υπάρχει ένα διμερές ε, πρόβλημα ανάμεσα στη Σλοβενία και την Κροατία. Ένα πρόβλημα που πρέπει να επιληθεί από τα ίδια τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί βέβαια να τίνει χείρα βοηθείας εφόσον συμφωνήσουν και τα δύο μέρη ε, τότε και εμείς ε, μπορούμε να βοηθήσουμε για να φτάσουμε πιο κοντά στη λύση. Βεβαίως ε, είναι σαφές ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να είναι πρόθυμες να επιδιώξουν το συμβιβασμό και να προβούν σε πραγματικές παραχωρήσεις. Αλλιώς ε, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζουμε στεναρά ότι το πρόβλημα αυτό που εμφανίστηκε κατά το παρελθόν δεν θα ε, μπλοκάρει την ένταξη των χωρών των ε, Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η σύγκρουση δεν είναι μόνο πρόβλημα για την Κροατία και τη Σλοβενία. Το πρόβλημα αυτό προκαλεί αλγινές αντιπώσεις ε, γενικότερα για το σύνολο της Ευρώπης και πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές γνωρίζουν ότι οφείλουν να επιδιώξουν τη λύση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν. Uh, concerning the energy policy, question of member of Europe, Szymanski. Uh, Κύριε Σιμάνσκι, για τα θέματα της ενέργειας, Όπως γνωρίζετε, ο αγωγός Ναμπούκο αυτή τη στιγμή είναι μια πρωτοβουλία που βρίσκεται στα χέρια ιδιωτικών εταιριών. Δεν ε, θίγονται άμεσα ή δεν συμμετέχουν άμεσα ευρωπαϊκές χώρες σε αυτόν τον, αυτό τον αγωγό. Πρέπει να βοηθήσουμε τις ιδιωτικές εταιρείες να ξεκινήσουν. Βεβαίως, εξακολουθεί να υφίσταται το θέμα του πώς θα η ικανοποιητική ποσότητα αερίου στον αγωγό Ναμπούκο. Πρέπει να ξεκινήσουμε ε, ουσιαστικό διάλογο με όλες τις άμεσα ενδιαφερόμενες χώρες και ως εκ τούτου η Τσεχία που είναι η προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανώνει μία ε, συνάντηση για τον αποκαλούμενο νότιο διάδρομο μία συνάντηση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ε, χώρες διαμετακόμισης όπως είναι η Τουρκία, η Γεωργία και η Αρμενία. Ε, αυτές θα είναι αφενός και από την άλλη πλευρά θα είναι όλες οι χώρες παραγωγή της Κασπίας θάλασσας. Νομίζω ότι αυτή θα είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση. Ως προς αυτά που είπε ο κύριος ε, Χόρατσεκ, θα ήθελα να σας πω προετοιμάζουμε μία συνάντηση Πρόκειται για μία συνάντηση όπου θα συζητηθούν θα συζητηθεί το ενδεχόμενο παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κύριε Τριανταφυλλίδη, ε, το θέμα με τον αγώνα Μπούκο νομίζω σας το εξήγησα ήδη. Σε τελική ανάλυση είναι προς όφελος της ε, Τουρκίας το να είναι μια αξιόπιστη χώρα διαμετακόμισης. Και θα ήταν προς όφελος της Τουρκίας να μην δώσω το κακό παράδειγμα. Το πετρέλαιο και το αέριο δεν μπορούν να γίνουν προαπαιτούμενα πολιτικών αποφάσεων. Η Τουρκία ως χώρα διαμετακόμισης ε, θα αποκομίσει μεγάλο κέρδος από ε, τη μεταφορά του αερίου και του πετρελαίου. Αυτό πρέπει να το πούμε, είναι σαφές. Όπως γνωρίζετε, η ε, Προεδρία της Τσεχίας είναι υπέρ του να ενταχθεί κάποια μέρα η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε ότι ε, θα υπάρξουν ε, μεταρρυθμίσεις ε, στην Τουρκία και από την άλλη πλευρά θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα λυθεί το πρόβλημα με την Κύπρο διότι αλλιώς βέβαια θα μπλοκαριστεί ο δρόμος ένταξης της Τουρκίας. Μισό λεπτό σχετικά ξέχασα να απαντήσω κάτι, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων. κατά πόσον ε, το γεγονός αυτό θα παραβιάσει, ε, θα επηρεάσει με συγχωρείτε τη συνεργασία μας με το Ισραήλ. Για να έχουμε καλές σχέσεις με το Ισραήλ πρέπει μέσα από το διάλογο να αποκομίσουμε και καλύτερη θέση για τους Παλαιστινίους. Όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται αποδεκτή ως πραγματικός εταίρος από το Ισραήλ, ε, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τίποτα σημαντικό. Τώρα οι Ισραηλινοί τουλάχιστον έχουν την ευήκονους ε, προς την πλευρά μας και αυτό αποτελεί μια επιτυχία της διπλωματίας. Βεβαίως θα μιλήσουμε ανοιχτά για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εφόσον παραβιεστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων ή οποιοδήποτε άλλου. Αλλά και πάλι σας λέω ότι είναι πραγματικά ε, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει τις ε, βέλτιστες δυνατές σχέσεις τόσο με τις αραβικές χώρες όσο και με το Ισραήλ. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Ο κύριος Πέτερλε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχήν να σας συγχαρώ για τους φιλόδοξους στόχους που θέσατε εκ μέρους της Τσεχικής Προεδρίας, ιδιαίτερος όσον αφορά την απόφαση να βοηθήσετε αυτές τις χώρες να χωρίσουν στο ΝΑΤΟ. Πιστεύω ότι η Προεδρία της Τσεχίας μπορεί να συμβάλλει ούτως ώστε να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις με την Κροατία και ελπίζω να αξιοποιήσει και η Κροατία μια, να, έχει, να έχει μια τεκμηρίωση για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ε, βεβαίως είναι το θέμα των συνόρων το οποίο η Κροατία θέτει στο προσκήνιο των συνομιλιών. Υπάρχει μια κοινή δήλωση του 1991 η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αρχή Πακτασού Σερβάντα. Μόνο με τον τρόπο αυτή, αυτό τόσο, θα βγουν ωφελημένες τόσο η Κροατία όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Σρότ έχει το λόγο. Συγγνώμη, ο κύριος Σρότ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε τρεις σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τη Λισαβόνα, γιατί είπατε ότι χρειαζόμαστε μια επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας, γιατί χρειαζόμαστε πιο συνεκτική πολιτική αμήνης. Και επίσης χρειαζόμαστε για την κοινή ενεργειακή πολιτική τη συνθήκη της Λισαβόνας. Όπως ε, ακούσατε από πολλούς ε, συναδέλφους, πολλοί θέτουν το ερώτημα για το πότε θα προβεί στην επικύρωση η δημοκρατία της Τσεχίας. Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα, πότε και κατά πόσο θα προβεί στην επικύρωση η Τσεχία. Δεύτερον, θα ήθελα να επανέλθω στη Γάζα. Είπατε ότι η δική μας ε, θέση του, η αντιμετώπιση του Ισραήλ δεν είναι πολύ ισχυρή. Δεν έχουμε συνομιλίες με τη Χαμάς. Έτσι λοιπόν πώ θα μπορέσουμε να οργανώσουμε όχι μόνο την ανθρωπιστική συνδρομή αλλά και τι ειρηνευτικές προσπάθειες. Πώ είναι δυνατόν να συμβάλλουμε στην διαδικασία ανοικοδόμηση, ή ανασυγκρότηση μάλλον στη Γάζα εάν δεν έχουμε καθόλου συνομιλίε με την χαμά, Είτε μα αρέσει η Χαμάς είτε όχι είναι γεγονό ότι η Γάζα διοικείται από τη χαμά. Η τρίτη μου ερώτηση έχει ω εξή. Συμφωνώ πλήρω με τι Προεδρίες τη τσεχική Προεδρία η, Τσεχία έχει πολλή εμπειρία όσον αφορά την, ε, τις ανατολικές χώρες και γειτονία με την Ανατολική Ευρώπη. Αλλά μιλάμε και για την ευρωμεσογειακή συνεργασία. Η Γαλλική Προεδρία νομίζω ότι πραγματικά έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα όσον αφορά αυτό το θέμα. Ε, ποιες είναι λοιπόν οι προτεραιότητε τη Τσεχία, τη Τσεχική προεδρία, όσον αφορά τη Μεσόγειο. Ο κύριος Ματσάκης έχει το λόγο. Κύριε ε, Υπουργέ, ε, συμφωνώ απολύτως όσον αφορά τις συνομιλίες με τη Χανάς, Χαμάς. Αλλά αν έχουμε έναν δημοκρατικό κατάλογο, γιατί εάν αποκηρύξει η Χαμάς ε, την τρομοκρατία θα βγει από το κατάλογο. Συνεπώς, ποια, είναι η λειτουργία αυτού του καταλόγου. Τώρα, όσον αφορά το ΝΑΤΟ, το, το ΝΑΤΟ είναι ο πυλώνας ασφάλειας της Ευρώπης και 26 από τα 27 μέλη είναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλη του ΝΑΤΟ, με μια εξαίρεση στην Κύπρο θα μπορέσετε να προσπαθήσετε να πείσετε την Κύπρο να κάνει αίτηση για προσχώρηση στο ΝΑΤΟ και θα προσπαθήσετε να πείσετε την Τουρκία να μην φέρει αντιδράση ή να, μάλλον να μην ασκήσει βέτο ε, σε σχέση με την προσχώρηση της Κύπρου. Τώρα, όσον αφορά τις καταστροφές στη Γάζα, πολλές από τις υποδομές εκεί έχουν καταστραφεί ολοσχερός και πολλές αυτές τις υποδομέ είχαν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς ε, θα λέγατε ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να πληρώσει για την ε, ανοικοδόμηση ή θα, και θα πρέπει η ΕΕ ή το Ισραήλ να πληρώσει για την ανασυγκρότηση. Τώρα, με τις αντιδράσεις από τη Ρωσία, με, το, με τους κινδύνους για την ειρήνη στην Ευρώπη, ε, τι γίνεται όσον αφορά την εγκατάσταση του αντιπυραυλικού συστήματος της Αμερικής στο έδαφος της Τσεχίας. Έχετε τώρα κάποιες αντιδράσεις σε αυτό ή όχι. Ή... Ο κύριος Πόσελτ. Ε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, εγώ είμαι εισηγητής για την Κροατία και το Κόσοβο, εκ του ΕΛΚ. Σκιώδης εισηγητής. Ε, θα ήθελα να πω το εξής ότι ανεξάρτητα από τη σχέση του διμερούς ζητήματος ποιες είναι οι δυνατότητες που βλέπετε να συμβάλλετε ούτως ώστε να ανοίξουν όλα τα κεφάλαια κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Τσεχίας. Κάτι το οποίο έχει απαιτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του να ολοκληρωθεί αυτό το έτος. Δεύτερον, η λύση για το κοσυφοπαίδιο βασίζεται στη πρόταση των Αβυσάρ ε, σεβασμός των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και το αδιέρετο του Κωσόβου. Τα δικαιώματα των μειονοτήτων είναι εδρεμένα στο Σύνταγμα του Κωσυφοπεδίου. Και η ΟΝΜΙΚ βρίσκεται υπό εξέλιξη. Αλλά τι γίνεται με το αδιέρετο του Κωσυφοπεδίου. Ε, επειδή η Ρωσία συμμετέχει στην ομάδα επαφής, ε, βλέπω ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι ως προς αυτό. Και ε, σε σχέση με σου είπε ο κ. βλέπετε κάποια δυνατότητα στο διάλογο με, το, με την ε, Ρωσία να μιλήσει. Απελευθερωθούν οι Κοτζακόφσκι και ο Λέμπεντεχ. Θα ήθελα να σας πω ότι η Τσεχία είναι μια χώρα της κεντρικής Ευρώπης και τώρα επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας εύχομαι λοιπόν ε, καλή επιτυχία και ελπίζω ότι θα έχετε σημαντικές πολιτικές επιτυχίες. Θα πρέπει να πω ότι με κατάπληξε την περασμένη εβδομάδα το Στρασβούργο κατά τη διάρκεια της συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ότι κανείς δεν ήταν παρόν εκ μέρους της Τσεχικής Προεδρίας ως παρατηρητής αυτή τη συζήτηση. Αυτό μου έκανε εντύπωση γιατί θυμούμε και πάλι τις παράνομες ε, συναντήσεις πριν από 20 χρόνια στα σύνορα με τη ε, Τσεχοσλοβακία στη Πολωνία, όταν ακριβώ τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούσαν μια σημαντική προτεραιότητα για μα ή κατά τη διάρκεια τη Γερμανική Προεδρία. Πάντοτε υπήρχαν παρατηρητέ σε αυτή τη ε, συνεδρίαση στο Στρασβούργο. Ε, πάντοτε υπήρχε ένα υπουργό αρμόδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτέ τι συζητήσει στο Στρασβούργο. Πώ εξηγείται λοιπόν αυτή την απουσία. Τώρα, όσον αφορά την ατζέντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Έχετε μια, κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα ε, σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, σε σχέση με τις ανησυχίες για τον αγωγό Ναμπούκο, το Κοινοβούλιο επεσήμανε το πόσο σημαντικό είναι να υπάρξουν και κάποιες οικονομικές δεσμεύσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία. Και θα ήθελα επίσης να αναφέρω αυτά τα οποία διαβάζουμε εδώ γνωμοδότηση του, στην τοποθέτηση του Μπαρόζο. Λέει ότι θέλουμε να έχουμε μια ταχεία συμφωνία στο Συμβούλιο ε, σε σχέση με τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ που δεν έχουν ταπανηθεί, τα οποία θα πρέπει να επενδυθούν στον τομέα της ενέργειας. Προτίθεται η Τσεχική Προεδρία λοιπόν να συστήσει να ακολουθήσουμε αυτή την πρόταση του Μπαρόζο. Και άλλη μια ερώτηση ε, σε σχέση με το πρόγραμμα του Μεντέντεφ για την επιδότηση ε, πριν από μερικούς μήνες για θέματα ασφαλείας. Φαίνεται ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή παγώνει αυτά τα προγράμματα. Ωστόσο το ζήτημα αυτό εκκρεμεί, παραμένει ανοιχτό. Τι πρόκειται να κάνετε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μπρόκ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω δύο σύντομες παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι η εξής. Είπατε ότι είσαστε σε στενή επαφή με την Ουάσιγκτον. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα η Αμερικανική κυβέρνηση το θέμα της Μέσης Ανατολής ε, να το ορίσει ως πρώτη προτεραιότητα έτσι ώστε να λυθούν και όλα τα προβλήματα μετά την εκεχηρία. Και θα ήθελα να σας στηρίξω σε αυτά που είπατε για τη Χαμάς. Η εταίροι μας είναι η μετριοπαθής ε, Παλαιστίνη ε, εκείνο που ενδιαφέρει είναι η απόσυρση των επίκων. Βεβαίω και δεν μπορούμε να συνομιλούμε με εκείνου που είναι τρομοκράτε, όπω πολύ σωστά είπατε. Το δεύτερο ερώτημα που θέτω αφορά στις δυσκολίε οι οποίες ε, αντιμετωπίστηκαν πολύ σωστά από την ε, τσοχική Προεδρία. Αναφέρομαι βέβαια στη συνθήκη της Λισαβόνας. Στο θέμα της ενέργειας λοιπόν δεν έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή έτσι ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία με τη Ρωσία έτσι ώστε ε, κάτω από αυτές τις συνθήκες να ε, εκμεταλλευτούμε τις ενοχές έτσι ώστε ή δυνατόν να διασφαλίσουμε την ενέργεια, να επιτύχουμε εγγυήσεις για την ενέργεια. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος του δεύτερου γύρου των συζητήσεων. Nicht mehr. bist du das hier? So, I would like to answer to member of the European Parliament. Uh, let's be quite open. Ας είμαστε ειλικρινείς. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να ενισχύσουμε να επιταχύνουμε την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τελικά η απόφαση είχε ληφθεί πριν από πολύ καιρό. Θα έπρεπε λοιπόν να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας αν η Κροατία πληρεί τις υποχρεώσεις της. Αλλά όπως σας είπα είναι σημαντικό να επιληθούν και τα διμερή προβλήματα με τη γειτονική της χώρα. Είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε, αλλά μόνο εφόσον το επιθυμούν και οι δύο πλευρές. Γιατί κατ' ουσίαν πρόκειται για ένα πρόβλημα που αφορά στις δύο πλευρές. Όσον αφορά τώρα στο θέμα που έθεξε ο κ. Ρότσεκ. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι όταν μιλάμε για την τσεχική επικύρωση, είναι σαν να μιλάμε για το θάνατο. Είμαι αρκετά αισιόδοξο ότι κάτι δύο θα γίνει στο εγγύς μέλλον, αλλά εγώ δεν είμαι μέλος του Κοινοβουλίου, γιατί στο Κοινοβούλιο αρέσει όταν ε, ορίζεται ένα χρονοδιάγραμμα σωστό είναι όταν τίθεται ένα χρονοδιάγραμμα να τηρείται. Είμαι αισιόδοξο. Η κύρωση ε, θα υπάρξει σύντομα. Είμαι σίγουρος ότι η Τσεχία θα επικυρώσει τη συνθήκη, αλλά δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή ε, ποια ημέρα ακριβώς. Όσον αφορά στη Γάζα, Είναι προφανές ότι η Χαμάς έχει πολύ ισχυρή θέση στη λωρίδα της Γάζας. Ε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Βεβαίως Το τι ακριβώς συμβαίνει στην ε, Γάζα δεν μπορούμε εμείς να ελέγξουμε τα πάντα, δεν μπορούμε να ελέγξουμε και τον απλό φορτωτή και φορτωτή. Εμείς πρέπει να μιλάμε με πολιτικούς όρους. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να έχουμε πολιτική συζήτηση με τη Χαμάς. Ε, έχουμε αφήσει εναποθέσει όλε όλες μας τις ελπίδες στην Αίγυπτο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στις επίσημες ε, επαφές της πρέπει να τηρεί τους κανόνες και να μην συνομιλεί με τρομοκρατικές οργανώσεις όσο δεν αποκηρύσουν τη βία. Και όχι μόνο λεκτικά, αλλά και επί της ουσίας. Ως προς την ανοικοδόμηση. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί το Φεβρουάριο ε, στο πλαίσιο μιας ε, συνεδρίασης και η Αίγυπτος είναι εκείνη ε, που θα επιληφθεί αυτής της συνάντησης. Η Αίγυπτος είναι εκείνη που έχει να λάβει τώρα τα της κατάπαυσης του πυρός καθότι συνορεύει με τη λωρίδα της Γάζας ζητήθηκε από την Αίγυπτο να οργανώσει αυτή τη συνάντηση και νομίζω ότι αυτό είναι και λογικό λόγω του ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας δεν είναι σημαντική μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ε, πολλές αραβικές χώρες που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Όσον αφορά τώρα στη Μεσογειακή Ένωση. Βεβαίως ε, θα συνεχίσουμε την πολιτική για τη Μεσογειακή Ένωση και η ανατολική εταιρική σχέση και αυτή είναι σημαντική, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού. Είμαστε σε στενή συνεργασία, ε, ξεκινήσαμε ουσιαστικούς διαλόγους με την Αίγυπτο, συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τη Γαλλία που βρίσκεται από την άλλη πλευρά της ε, Μεσογείου ε, και νομίζω ότι ανάλογα με τις ε, συνθήκες οι οποίες μετά τη σύγκρουση κατέστησαν πιο δύσκολες αυτό το δέχομαι και συμφωνώ αλλά νομίζω ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πρόοδο και στο θέμα της Μεσογειακής Ένωσης. Τώρα, όσον αφορά τη Χαμάς και τον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων. Σας είπα, το θέμα δεν είναι μόνο ε, λεκτικά να αποκηρύξει η Χαμάς ε, τη βία. Το θέμα είναι να ε, μην καταφεύγει πλέον σε τρομοκρατικές ενέργειες. Είδαμε ότι στην Ιρλανδία, παραδείγματο χάρη, σημειώθηκε επιτυχία. Ο ένοπλος ε, στρατός ε, είπε ότι ε, δεν θα προβαίνει πλέον σε ένοπλες επιθέσεις. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έπαυσαν οι ένοπλες επιθέσεις έπαυσαν οι τρομοκρατικές ενέργειες, άρα τους διαγράψαμε από τον ε, τρομοκρατικό κατάλογο. Περίπου το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για τη Όσον αφορά τώρα στο ΝΑΤΟ. Βεβαίως μέλος του ΝΑΤΟ μπορεί κανείς να καταστεί μόνο εφόσον όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ε, συμφωνήσουν επ' αυτού. Δηλαδή ε, πρέπει όλα τα κράτη, αν όλοι συμφωνούσαν ε, ε, για να καταστεί ένα κράτος μέλος, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα από αυτού. Όσον αφορά στην υποδομή στη Γάζα, Δεν ξέρω τι θα γίνει και με τι Ηνωμένε Πολιτείε, τι θα κάνουν και αυτές, ε, κατά πόσον θα βοηθήσουν, τι θα κάνει και το Ισραήλ. Πιστεύω όμως ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανοικοδόμησης ε, θα δοθεί ε, από τις αραβικές χώρες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι πρέπει και εγώ να ομολογήσω ότι είναι ενοχλητικό το να πρέπει κανεί να αποκαθιστά συνεχώ το κτίριο που ε, καταστρέφεται και έχει και το παρελθόν πολλές φορές. Επειδή όμως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλούσια περιοχή, δεν μπορούμε να πούμε όχι σε όσους έχουν την ανάγκη μας. Και οι άνθρωποι που βρίσκονται στη Γάζα έχουν πραγματικά την ανάγκη μας. Έτσι λοιπόν, ε, παρά την ενόχληση που αισθανόμεθα όλοι μας, θα πρέπει να τους βοηθήσουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πόσελτ κάτι, να απευθυνθώ σε αυτόν. Κοιτάξτε, όσον αφορά την ε, Κροατία, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανοίξουν τα κεφάλαια που είναι απαραίτητο να συμβεί αυτό ε, για την ένταξη της Κροατίας. Βεβαίως ε, θέλουμε να πούμε ότι αυτή δεν είναι η μόνη περίπτωση όπου μπλοκαρίστηκε η διαδικασία της ένταξης. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά και η Κύπρος ε, μπλοκάρισε την ε, ένταξη της ε, Τουρκίας. Το κακό παράδειγμα, πολλοί είναι πρόθυμοι να το ακολουθήσουν, άρα δηλαδή βλέπουμε το ίδιο συμβαίνει τώρα και με την Κροατία. Πάμε στο Κωσυφοπέδιο. Βεβαίως και από αυτού είναι ενιαίο το κεσοπέδιο έχουμε πει και είναι αδιέρετο επίσης ε, αυτός ο ισχυρισμό ε, ευσταθεί και βεβαίω όμως θεωρώ ότι για κάποιο χρονικό διαστήμα θα πρέπει να αποδεχθούμε την κατάσταση όσο έχει. Θα πρέπει επίσης να αντισταθούμε στον πειρασμό του να θέλουμε να επιβάλλουμε την άποψή μας. Βεβαίω, από την άλλη μεριά, έχει αλλάξει το σκηνικό στην Σερβία. Και θα πρέπει να αποδεχθούμε την κατάσταση όσο έχει. και βεβαίω η βία έλαβε χώρα εκεί και ε, οι δύο πλευρές οφείλονται ευθύνονται συγγνώμη θα πρέπει όμως να δεχθούμε ότι κατά μία μεταβλητική περίοδο τα πράγματα θα τα δεχθούμε ως έχουν και ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι δυνατόν να υπάρξει μια διοίκηση θα προχωρήσουμε βήμα-βήμα. Yeah, Επίση. Ε, that Ίσως δεν πρέπει να είμαστε εκεί όταν συζητήθηκε η υπόθεση των δικαιωμάτων στο Στασβούργο. Όπως γνωρίζετε, πάντως αποτελεί προτεραιότητα της Προεδρίας μας. Όντως. Η αλήθεια είναι ότι Ε, είχαμε διμέτωπο ούτως είπε αγώνα το φυσικό αέριο και από την άλλη την προϊόντα της Γάζας και γι' αυτό και δεν είναι παρέστημενη στην συζήτηση υποθέσεις του Στρασβούργου πάντως ελπίζουμε ότι θα εκπροσωπηθούμε βιώντας την επόμενη συζήτηση επίσης ε, θα καταβληθεί πάσα προσπάθεια να γίνει αυτό το οποίο είπαμε διότι, διότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, είναι πολύ ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων Τώρα στρατηγική για την τήρηση των δικαιωμάτων που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να επιμείνουμε να μιλήσουμε με όλους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα πρέπει να τονιστεί προς όλες κατευθύνσεις ότι πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικό στοιχειώδες πρωτής σημασία θέμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκάθαρες απόψεις να είναι μια παρένθεση κάθε αυλεψία κατά την οποία δεν προσέχουμε διόντες τα δικαιώματα. Αυτό θα πρέπει επομένως να το τονίσουμε στους ε, εταίρους μας όλους προς πάσα κατεύθυνση. Και προς όλους εκείνους οι οποίοι τα έχουν παραμελήσει τελείως on our uh, policy of human rights. We are supporting human rights movements and uh, and, NGOs uh, all over the world. Γι' αυτό και θέλουμε να συνεργαστούμε, να υποστηρίξουμε τα, τα κινήματα, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, πα, πα, πάντα φορέα όσο έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκτός βέβαια και σε Κούβα, σε Ρωσία, σε, σε, σε, σε, σε Βυρμανία, παντού. Ελπίζω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημορφωθεί μια νέα πολιτική για δημοκρατία και δημοκρατισμό και ανθρώπινα δικαιώματα που και ελπίζουμε ότι αυτό μας το πρόγραμμα εργασίας θα γίνει αποδεκτό φέτος κιόλας. για τον αγώνα Ναμπούκο ήδη μίλησαμε. Αν δεν δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό θα πρόκειται για πολύ σημαντικό επίτευγμα και εμείς θα βοηθήσουμε κάθε προσπάθεια κάθε προσπάθεια εκταμίευσης πόρων ούτως ώστε να υπάρξει η κατάλληλη υποδομή γιατί ακριβώς το ενεργειακό είναι πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικό ε, θέμα είναι τρομερή μας ε, ε, παράληψη ότι δεν έχουμε διαμορφωσμένη κοινή πολιτική για την ενέργεια και μόνο σε συνεργασία με την Κομισιόν θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εκταμιεύσουμε τους απαραίτητους πόρους για να υπάρξουν κατελέσεις επενδύσεις ε, Επίσης παρακολουθώ να αναφέρθηκε ότι κάποια στιγμή μέσα στην κρίση το περίφημο σχέδιο μας δεν πέφτουν αμενόμενα κάποια μέρα θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα με με δεδομένα το πώς διαμορφώνεται η στάση της Ρωσίας, της νέας Ρωσίας, αν και δεν είναι τόσο νέα αυτά. Αυτά υπάρχουν εδώ και δεκαετίες από τη Σοβιετική Ένωση, τα ξέρει εδώ καλά ο Πολωνός φίλος. Το σχέδιο Ραπάτσκι, ε, τώρα πάντως δεν, δεν ξέρω είναι με τον πρόεδρο Μέντιο δεν ήταν και τόσο έτοιμος μάλλον έτσι έριχνε ιδέες στο τραπέζι πάντως σε επαφές με τους Ρώσους θα πρέπει να προσέξουμε θα συνεχίσουμε τις επαφές θεωρώ πάντως ότι η αρχιτεκτονική ασφάλεια είναι καλή στην Ευρώπη και θα ήταν ακόμα καλύτερη εάν όλοι όλοι συμμορφώνονται Οπότε, αν τηρήσουν τα επεσχημένα και οι Ρώσοι, θα αποκτήσουν περισσότερη αξιοπιστία. Με δεδομένη λοιπόν τέτοιου είδους πρόοδο, τότε μπορούμε να κάτσουμε να συζητήσουμε κάποια καινούργια θέματα, αλλά προς το παρόν η πολιτική που μπορούμε να ακολουθήσουμε είναι αυτή εν ώψη νέας πολιτικής, νέας δομής των πραγμάτων. Μια που είδαμε τι γίνεται σε περιόδους και στιγμές κρίσης, ότι έχουμε εμπλοκή στον υπάρχοντα μηχανισμό. Άρα να προσέξουμε και να δούμε κατά πόσο χρειάζεται κάτι καινούριο στον υπάρχοντα παλιό μηχανισμό ασφάλειας. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, λέει ο και τώρα πάμε τρίτο. Α, μισό λεπτό κάτι ξέχασα λέει ο κύριος Σβάρτζεμπεργκ. Ξεχάσα τον κύριο πρόγραμμα. Πώς τολμήσατε λέει ο πρόεδρος. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Τον ξέρω τον κύριο Έλμαρ Μπρόκ. Δεν ξέρω τι πιστεύει σε σχέση με κάποιες τύψεις που αισθάνονται οι Ρώσοι. Εγώ τέτοιο πράγμα δεν το καταλαβαίνω αντιθέτω. Αντιθέτω, μια χαρά είναι. Ενθουσιασμένοι είναι εκεί πέρα. We όμω, όμως και θα πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι, να μιλήσουμε με τους Ρώσους, να γίνει διάλογος εντατικός. ελπίζοντας ότι κάτι θα βγει. Τα πράγματα προς το παρόν πάντως είναι δύσκολα. Αλλά προ το παρόν αυτό δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μα. Άλλη στρατηγική δεν υπάρχει για να αποσπάσουν τίποτα άλλο τη Ρωσία. Τα θυμάμαι και από τα νιάτα μου αυτά. Θυμάμαι τον κύριο Γκρομίκο που ήταν διαβόητος για το νιέτ, το όχι πολύ. Πάντως αυτή τη φορά ελπίζω κάτι να αποσπάσουμε. Όχι επειδή έχουν νιώθουν τύψεις, αλλά ίσως επειδή θα συνειδητοποιήσουν. ότι από την προστριβή τους με την Ουκρανία εμείς πλώσαμε την ίδια. Και εκείνοι, οι Ρώσοι, έχασαν σε φήμη και αξιοπιστία. Προσωπικά, πιστεύω ότι η σχέση μας με τη Ρωσία είναι πάρα πολύ βασικό ζήτημα. Και θα πρέπει να γίνει αντικείμενο μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής. βλέπουμε από μια μεριά την τάση κάποιοι νέοι πολιτικοί να αναγιοποιούν το Κρεμλίνο. Ελπίζοντας ότι κάτι θα αποσπάσουν. Και το σύνολο πάντως Ευρώπης ποτέ δεν θα φέρει με αυτόν τον τρόπο. αν δεν βρει μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Thank you, thank you, uh, uh... Minister, for two things. First, that you did not omit Elmar Second... Uh, Ευχαριστούμε πρώτα πρώτα που απαντήσατε στον Μπροκ. Λέει ο Πρόεδρος από την άλλη. Ξέρουμε ότι έχετε μακρά μνήμη, έχετε πολλές κανένα αναμνήσεις για την εξωτερική πολιτική στην Ανατολική Ευρώπη και χρειάζεται αυτό για να μην επαναλαμβάνεται η ιστορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα προχωρούμε στον τελευταίο γύρο. Εδώ θα είμαι ακόμα πιο αυστήρο, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχετε. Πόση ώρα έχετε, όσο θέλετε, αμάν λέει. Αλλή μονό μας λέει ο πρόεδρο. Πάνε ψηφοφορία. Οπότε, το πολύ ένα λεπτό και θα είμαι πανάυστηρος. Χιμπάσκοβα. Χιμπάσκοπα. ορίσατε πρόεδρε. Πρώτα πρώτα σας ευχαριστώ για τις προσπάθειές σας, για την ε, Γάζα και δεύτερον σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Είμαι σίγουρος ότι όχι μόνο η δική μας χώρα, αλλά το σύνολο της Ευρώπης χρειάζεται My is... αυτή την, την συνθήκη. Τώρα όσον αφορά τη συνθήκη στη Γάζα, συχνά μας αναφέρετε στην εισηγησή σας, το Ιράν, και τις άλλες χώρες εκεί. Τι γίνεται εκεί πέρα, ε, πώς, πώς ε, θα αντικοτουρίζεται η πολιτική μας ε, για τη Γάζα σε σχέση με την πολιτική μας για την Συρία με σχέσεις τώρα. Θεωρώ ότι ακρογωνίας λίθος στο μέλλον για μεσοπρόθεσμη διαμόρφωση αυτής της πολιτικής θα είναι το τι θα κάνουμε για το Αφγανιστάν. Εδώ δεν είμαστε το ΝΑΤΟ, το ξέρω. Όμως το πρώτη της Ένωσης προς το Αφγανιστάν. Τρίτη ερώτηση. Την κόβει ο Πρόεδρος και δεν ακούγεται η ομιλήτρια. You've asked us two questions. Sorry. Sorry. Uh, now we pass to Mm, signora Napoletano, prego. Grazie Presidente. Io non voglio... Ναπολιτάνο, εγώ δεν θέλω να επασπώ κανένα, θέλω να σας πενθυμίσω ότι ε, ε, με αυτή την κίνηση θέλαμε να υπάρξει μια μαγδά αναχώρηση αλλά δεν έγινε τίποτα παρέμεινε το εμπάργο στην ε, Γάζα γι' αυτό και εγώ σας λέω προσέξτε θα πρέπει το να μπούμε μας να τον αναγκάσουμε να να υποχωρήσει έτσι θα αποδυναμωθεί η στάση του άρα η ανοικοδόμηση δεν θα πρέπει να γίνεται φορτισμένη ε, συναισθηματικά, ιδεολογικά μην ακούγεται μόνο το Ισραήλ, μόνο το Σαρκοζή ας κάτσουμε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά τους Παλαιστινίους η Δένωση για την Μεσόγειο μια που ήδη και για αυτό το θέμα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή είναι τέτοιο που θα πρέπει ο Σαρκοζή να αποκτήσει την ευκαιρία να συνεχίσει με τον Μπάρκ να είναι συμπρόεδρος μέχρι ότου η συνθήκη της Λισαβόνας τεθεί σε ισχύ. Duff. Uh, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της τρομοκρατίας. Οι Βρετανοί άρχισαν να, μιλούν, να συνομιλούν με τους Ιρλανδούς πριν να σταματήσει ο Ήρα να σκοτώνει τους ανθρώπους αλλά το ερώτημά μου αναφέρει τα στρατεύματα τα οποία θα αναπτύξουν οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και οι Βρετανοί στα σύνορα της Γάζας. Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι τρεις αυτές χώρες πρόκειται να αναπτύξουν στρατεύματα στην Παλαιστίνη, έστω για κάποιο διάστημα. Και θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ θα εκτιμούσα πάρα πολύ να μας πείτε αν μας λέγατε κάποια πράγματα για το μέγεθος των στρατευμάτων, το, τη διάρκεια παραμονής τους, τους, τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν κλπ. Κύριε Σουάρτσενμπεργκ, μπορείτε να μας υποσχεθείτε ότι θα ενημερωθεί το Κοινοβούλιο και θα συμμετέχει στη διαβούλευση σε σχέση με την ανάπτυξη αυτών των ε, ομάδων, των στρατευμάτων της αποστολής αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γκάλερ έχει το λόγο. Ναι, σας εύχομαι κάθε επιτυχία για την Προεδρία σας. Δεν βλέπετε ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν ε, κοινέ ε, θέσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, νομίζω ότι ίσως θα μπορούσαμε να το πετύχουμε σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, ούτως ώστε να υπάρχει μια κοινή στάση εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας σε σχέση με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Δεύτερον, σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριος Ντάφ, θα πρέπει να πω ότι έχω την ανησυχία ότι τώρα ναι, μεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, θα προβούμε στην ανασυγκρότηση, αλλά δεν υπάρχει δεδηλωμένη βούληση να υπάρχει μια στεναρή παρουσία στην περιοχή αυτή ούτως ώστε πραγματικά να καταστήσουμε σαφή, ξεκάθαρη τη δέσμευσή μας εκεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Η κυρία Κόμες, κύριε Υπουργέ, στο κεφάλαιο των διατλαντικών σχέσεων, μία από τις προτεραιότητες που έθεσε ο κύριος Ομπάμα είναι ότι θέλει να κλείσει το Γκουαντάναμο και όλο αυτό το μοντέλο με μεταφορά της σε μια άλλη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει μια συντονισμένη προσέγγιση σε σχέση με το Γκουαντάναμο. Αλλά πού βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία; μπορείτε να μας πείτε κύριε Υπουργέ. Το Γκουαντάναμο θα είναι ένα βασικό σημείο σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Και ε, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής μια συγκεκριμένη στρατηγική. Ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος ε, Λαντσμπέργκης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, ο ατέρμον πόλεμος στην ε, Παλαιστίνη δεν θα πάρει ποτέ ένα τέλος. Κατά την άποψή σας, εάν οι Ισραηλοί δεν πάρουν πάλι το δρόμο της εξορίας ή αν η Χαμάς δεν αλλάξει γνώμη, η Χαμάς και το Ιράν θα ήθελα να προσθέσω. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι σαφές για όλους έστω και αν υπάρχει μια αλλαγή φρονήματος εκ μέρους της Χαμάς. Θα δώσει η Χαμάς ποτέ την προτεραιότητα στην ειρήνη σε σχέση με τον πόλεμο. Η προτίθεται η Χαμάς να συνεργαστεί με το Ισραήλ παρά να συνεχίζει τις καταστροφές. Οι πύραυλοι κατά του... Με τους πυράβλους κατά του Ιράν τι θα γίνει. Νομίζω αυτές είναι οι ερωτήσεις που θα έπρεπε να θέσει κανείς προς τη Χαμάς ίσως θα μπορούσαμε με τον τρόπο αυτό να έχουμε μία μικρή διευκρίνηση των πραγματικών του στόχων. Η Παλαιστίνη ασφαλώς υποφέρει τα πάνδυνα και είναι η κατάλληλη στιγμή να διατυπώσουμε μία έκκληση για να τους πούμε να αλλάξουν στάση. Αλλά νομίζω ότι αυτό εγκυμονεί τον κίνδυνο να προκαλέσει την θυμηδία της παγκοσμίου κοινότητας. Παρ' όλα αυτά αξίζει τον κόπο. Ο κύριος Κύριε Υπουργέ, ε, δεν νομίζω ότι απαντήσατε στον προηγούμενο γύρο στην ερώτηση του συναδέλφου από την Κύπρο. Η δική ε, και η ερώτηση που θα ήθελα να σας απευθύνω είναι πώς αντιμετωπίσετε τη σχέση με τη Ρωσία δεν μπορούν να βελτιωθούν οι σχέσεις αυτές με τη Ρωσία μέσω μιας ε, βελτιωμένης ατμόσφαιρας εδώ με το να αποστασιοποιηθεί κανείς από την πρόθεση εγκατάστασης του αντιπυραυλικού συστήματος των ΙΠΑ στην ε, Τσεχία. Και σας ε, ρωτώ σαν εκπρόσωπο μιας χώρας που συμμετέχει σε κάτι τέτοιο. Ξέρουμε ότι η Ρωσία θεωρεί ότι αποτελεί ένα κίνδυνο για τα δικά της ε, προγράμματα. Ε, και νομίζω ότι θα οδηγήσει σε μια νέα κλιμάκωση των εξοπλισμών. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σε σχέση με τον υπόθηκε ότι αν η Κομισιόν ξεπαγώσει κάποια κονδύλια Ίσως αυτό θα ήταν ε, μια καλή ιδέα. Δεν έχουμε ένα εκπρόσωπο της Κομισιόν εδώ. Ε, θα προβεί σε αυτό το ξεπάγωμα των κοντιλίων η Κομισιόν, δεν ξέρω, μπορείτε να μας πείτε εσείς. Ε, δεν ξέρουμε ποια είναι η στάση της Κομισιόν. Τώρα, όσον αφορά την Τρόικα, η Γαλλική και η Σουηδική Προεδρία, οι προηγούμενες Προεδρίες βρίσκονται σε διαβούλευση μαζί του ιδιαίτερα όσον αφορά τη στρατηγική της Βαλτική για την, Ευρωπα... για την Μεσόγειο και την Βαλτική. Όταν οι Βρετανοί είχαν μια, θητή, είχαν μια εντολή στην Παλαιστίνη, οι μέλη της δικής μου οικογένειας είχαν στυλιτευτεί ως τρομοκράτες. Δεν ξέρω, ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε πιο πολύ εις βάθος και να σκεφτούμε κατά πόσο δεν θα συγκαλέσατε μία συνεδρίαση στην Πράγα μετά την, ε, τις εκλογές στο Ισραήλ μαζί με τις Ηνωμένε Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ ούτως ώστε να μην απομακρυνθούμε υπερβολικά πολύ από τις συμφωνίες του Καμπ Ντέιβιτ. Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο. important Λοιπόν, ε, θα πρέπει να θέσουμε το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της ε, πολιτικής κατάστασης ε, ιδιαίτερο στην Γάζα και σε όλη την Παλαιστίνη. Όπως ξέρετε υπάρχουν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες που προσπαθούν να κάνουν κάποιες συνομιλίες όπως ο Γερμανός Υπουργός και ο πρόεδρος κ. Σαρκοζή ο οποίος προσπάθησε να συνομιλήσει με τους Σύριους, με τη Συρία και πήγε στην Δαμασκό με το σκοπό αυτό. Φαίνεται το αποτέλεσμα ήταν ότι η Συρία είπε ναι στην κατάπαυση του πυρός γιατί φαίνεται ότι όχι μόνο η Χαμάς, ε, ε, όχι, ότι η ίδια ηγεσία της Χαμάς, η οποία έχει την έδρα της στην ε, Δαμασκό, αποδέχτηκε την κατάπαυση του πυρός. Όχι μόνο οι αγωνιστές της Χαμάς. Δηλαδή υπήρξαν κάποια αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης. Τώρα, όσον αφορά το Ιράν, Δεν υπάρχει αφιβολία ότι τη βασική χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της ε, Χαμάς και της Χεσμολάχ προέρχεται από το Ιράν. Αυτό νομίζω είναι αρκετά προφανές. Και βεβαίως έχουν σημαντική επιρροή. Γίνονται συζητήσεις μεταξύ του Ιράν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων πολιτιών. Η θέση του Ιράν ε, ωστόσο μέχρι στιγμής ε, δεν αλλάζει. Το Αφγανιστάν συμμετείχε σε μια συνάντηση κορυφής μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. η πρόσπιση της δημοκρατίας ε, στο Αφγανιστάν βεβαίως αποτελεί πρωτίστως μέλημα του ΝΑΤΟ, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικές είναι οι δικές μας προσπάθειες στο Αφγανιστάν παρόλα αυτά. Ε, και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη, καθώς και οι επιμέρους χώρες μέλη θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα πράγματα γιατί τελικά είναι οι δικέ μας ελευθερίες που διακυβεύονται και η δική μας ασφάλεια που διακυβεύονται στο Αφγανιστάν και που τις υπερασπιζόμαστε εκεί και θα πρέπει να το έχουμε αυτό πάντοτε κατά νου. Η κυρία Ναπολιτάνο, κυρία Ναπολιτάνο, πιστεύω ότι είναι μείζονος σημασίας να ενισχύσουμε τη θέση του Πρόεδρου Αμπάς. Όχι μόνο στα κατεχόμενα εδάφη, αλλά και στη λωρίδα της Γάζας. Νομίζω ότι αυτό είναι τεράστια σημασία. Η Χαμάς, όπως σας είπα, όσο εμένει στους ε, τρομοκρατικούς της σκοπούς δεν μπορεί να είναι επίσημος εταίρος της της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε ότι ασκεί σημαντική επιρροή στη λωρίδα της Γάζας και υπάρχουν Uh, Και όποιος ε, δουλεύει, έχει επαφές στην, ε, ε, στη λωρίδα της Γάζας, έχει κάποιες επαφές με τη Χαμάς. Τώρα, η ανασυγκρότηση. Θα συζητηθεί βεβαίως στη συνδιάσκεψη που έχει προγραμματιστεί το Φεβρουάριο από την Αίγυπτο. Και βεβαίως ε, θα παραστούμε και εμείς εκεί και ε, στοχεύουμε σε σημαντικά αποτελέσματα. Όσον αφορά τη Μεσογειακή Ένωση, πιστεύω ότι βρήκαμε μια πολύ καλή λύση με τη Γαλλική Προεδρία, μια λύση η οποία λειτουργεί καλά και όπου ο ρόλος της Γαλλίας και του Προέδρου κ. Σαρκοζή εκπληρώνει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκε μια προσέγγιση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου και δεν υπάρχει το θέμα της του ποιος προεδρεύει και πώς. Το ερώτημα τώρα του κυρίου Νταφ ε, σε σχέση με τον Ήρα. Ξέρω πώς συνέβησαν τα πράγματα. Αλλά υπήρξε μια επίσημη, ε, υπήρξαν επίσημες συζητήσεις μεταξύ της Βρετανικής κυβέρνησης και του Ήρα. Αλλά εγώ υπήρξαν ανεπίσημες συζητήσεις, αλλά εγώ τώρα ε, μιλάω για επίσημες επαφές όταν αναφέρομαι στη Χαμάς. Μιλώ για επίσημες επαφές. Μπορούμε να έχουμε κάποιες άτυπες επαφές, αλλά δεν είναι δυνατόν. να έχουμε επίσημες επαφές. Τώρα, όσον αφορά τον ε, τετραμερή διάλογο, νομίζω ότι κάθε πλευρά προσπαθεί για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Το κουαρτέτο θα συνέλθει μάλλον το Μάιο. Ενδεχομένως θα υπάρξει προηγουμένως μία προπαρασκευαστική συνάντηση λόγω ακριβώς της κατεπίγουσας φύσης της ε, κατάστασης. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα αρκετά χρήσιμο εργαλείο ένα ακόμα επιπλέον εργαλείο εκτός από τα πολλά διπλωματικά εργαλεία που υπάρχουν την επίλυση των προβλημάτων εκεί. Δεν έχουμε ευρωπαϊκά στρατεύματα ή πλοία στην περιοχή. Ε, έγιναν εξεγγλίες από ορισμένε χώρες όπως είναι η πλοια στην περιοχη εγιναν εξεγγλιες απο ορισμενε χωρες οπως ειναι η Ισπανία, ίσως η Γερμανία, δεν ξέρω. και έγινε μια έκκληση εκ μέρους των χωρών αυτών να βοηθηθούν οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της Γάζας. Δεν είναι λοιπόν μια αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα θέμα που αφορά την κάθε κυβέρνηση ξεχωριστά και θα πρέπει να διεξαχθεί η συζήτηση σε εθνικό επίπεδο εκ μέρους της κάθε χώρας κατά πόσο επιθυμεί να αποστείλει βοήθεια. Τώρα όσον αφορά το Γκουαντάναμο, βεβαίως είναι κατεπήγον ε, το ζήτημα αυτό. Ε, είναι κυβέρνηση της Αμερικής έχει κατ' επανάληψη δεσμευθεί να κλείσει το Γκουαντάναμο, αυτό το φρικιαστικό μέρος. Βεβαίως ε, τίθεται το θέμα το τι θα γίνουν οι φυλακισμένοι του Γκουαντάναμο. Κατά πόσο θα ζητηθεί από κάποιες χώρες της Ευρώπης ή την Αυστραλία να αποδεχθούν τους πρώην κρατούμενους του Γκουαντάναμο. Νομίζω ότι θα έπρεπε πρώτα να ρωτήσουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε πώς από αυτούς τους κρατούμενους ε, προτίθενται να δεχθούν ήδη και στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αλλά δεν είναι δικό μου θέμα να επιλύσω αυτό το πρόβλημα. Εγώ δεν θα απαγορεύσω σε καμία ευρωπαϊκή χώρα να δεχτεί αυτή την αμερικανική, το αμερικανικό αίτημα. MEP Όσον αφορά τους πυράβλους, κύριε σε εσάς απευθύνομαι. όσον αφορά περισσότερο ε, στην ε, αντιπυραυλική ασπίδα ε, που προστατεύει την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Εδώ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η ασπίδα προστατεύει και την Ευρώπη. Γιατί αν τη δείτε τελικά να κατασκευάζεται θα δείτε ότι προστατεύει την Ευρώπη. Με αυτή την αντιπυραυλική σπίδα κατορθώσαμε να την εντάξουμε στο ΝΑΤΟ και αυτός ήταν ε, ο πρωταρχικός στόχος της ε, διπλωματίας μας. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ επιτύχαμε το στόχο μας. Ε, ξέρω ότι υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από πλευράς της Ρωσίας, στρατηγοί και άλλοι Ρώσοι λένε ότι θα στρέψουν και εκείνοι τους ε, πυράβλους τους ε, προς την ε, Τσεχία αν κατασκευαστεί αυτή η ασπίδα. Εμείς βέβαια θα έχουμε μόνο τα ραντάρ. Έχω τη χαρά να σας πω ότι το σύστημα αυτό δεν στρέφεται κατά της Ρωσίας, ούτε τα ραντάρ ούτε οι πύραυλοι που θα εγκατασταθούν στην Πολωνία. Ο μόνος στόχος είναι με κινητική ενέργεια να ε, εξουδετερώσουν εχθρικούς ε, πυράβλους που ενδέχεται να εκτοξευθούν. Ε, βέβαια για να το συζητήσουμε πρέπει να γνωρίζουμε και όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες. Είναι θέμα αμυνάς μας ε, για το μέλλον και πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι αρκετές χώρες στην Ανατολική και την Νότιο Ανατολική Ασία ήδη τώρα έχουν στη διάθεσή τους πυρηνικά όπλα ή προετοιμάζονται για να τα αποκτήσουν. Ενώ εμείς ε, προετοιμαζόμεθα για πυράβλους ε, μικρούς και μεγάλου ελληνικούς. Όλα αυτά για το μέλλον. Επειδή λοιπόν ε, υπάρχουν κάποια καθεστώτα ε, που δημιουργούν κάποια προβλήματα, καλύτερα να προετοιμαστούμε έγκαιρα. Πιστεύουμε ότι ο κίνδυνος δεν, δεν υπάρχει σήμερα, αλλά ε, ίσως μετά από 10 χρόνια. Και ε, μέχρι τότε βέβαια το σύστημα θα είναι έτοιμο, θα έχει εγκατασταθεί το ραντάρ στην τσεχική δημοκρατία. και πριν γίνει η εγκατάσταση των πυράβλων στην ε, Πολωνία θα περάσουν πολλά χρόνια. Ε, όλα αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί ε, κατά το 2020. Νομίζω λοιπόν ότι ένα παρεμφερές ραντάρ υπάρχει ήδη στο Λέτι Σόιλ και στο Ντάνι τη Δανία και τη Μεγάλη Βρετανία. Και οι δύο αυτές χώρες δεν συζήτησαν αυτό το θέμα με άλλους ε, ευρωπαϊκούς εταίρους. Εγκατέστησαν αυτά τα συστήματα μετά από δική τους και μόνο απόφαση. Αυτό κάναμε και εμείς. σε είναι σημαντικά στοιχεία για την ε, άμυνα της Ευρώπης ε, στο μέλλον και σας παρακαλώ να τα δεχτείτε αυτά ε, ως τέτοια. Κύριε Υπουργέ, καλύψατε... Μισό λεπτό. Ξεχάσατε μήπως κάτι. δεν ξέρω αν πρέπει εγώ να απαντήσω στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εσείς μήπως καλύτερα, εμείς απλά προεδρεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως να πω ότι ε, θα υπάρξουν διαβουλεύσεις ε, στο μέλλον το να υπάρξει μια ε, συνδιάσκεψη στην Πράγα για το θέμα της Μέσης Ανατολής θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αν τελικά ε, διαρκέσει η ειρηνευτική διαδικασία. Και ε, θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα της συνάντησης και πώς θα εμπλακεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας από τους ε, στόχους της επίσκεψής μου στη Ρωσία τον επόμενο μήνα είναι ακριβώς να αρχίσω ε, διαπραγματεύσεις ε, με την Αμερικανική κυβέρνηση έτσι ώστε να μην κάνουν τα ίδια λάθη που έκανε και ο Κλίντον και ο κύριος Μπούς που μετέθεσαν το πρόβλημα της ε, Μέσης Ανατολής ε, στο τέλος του καταλόγου των προτεραιοτήτων τους. Θα πρέπει η κυβέρνηση να γνωρίζει ότι ε, το θέμα επίγει. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Βεβαίως σας κάναμε ερωτήσεις που αφορούν επί του επιστήτου. Ελπίζουμε έστω να, να μπορέσετε να συμβάλλετε στο να επιληθούν και στα μισά και σας ευχόμεθα κάθε καλό κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Ματιός. No. So, colleagues, we still have some work to do this afternoon. Συνάδελφοι, ε, πρέπει να συνεχίσουμε. Θα ξεκινήσουμε με το σημείο 17 ετήσια έκθεση σχετικά με τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΑ. Ο εισηγητής είναι ο πρόεδρός μας, ο Τζάζεκ Σάριος Βόλσκι και θα του δώσω το λόγο. Λοιπόν, η έκθεση συνιστά μια ετήσια προσπάθεια και να έχουμε ένα διάλογο με το Συμβούλιο για την ΚΕΠΑ και προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα κάπως πιο διαφορετικά θέτοντας ε, περισσότερα αιτήματα στην πλευρά του Συμβουλίου και ε, προσπαθώντας να κάνουμε πιο εστιασμένοι, ε, πιο επικεντρωμένοι στους στόχους μας και λιγότερο περιγραφικοί γιατί το Συμβούλιο συνήθως ε, καταρτίζει ένα απλό κατάλογο αν εμείς θέλουμε να έχει έναν περισσότερο στρατηγικό χαρακτήρα. Η έκθεση αυτή ε, ασχολείται στη δεύτερη εκδοχή με τα περισσότερα ε, περισσότερες από τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και τελικά προτείνει 14 ε, συμβιβασμούς. Δεν ξέρω αν κάτι έχει παραλυφθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με αυτές τις απόψεις, αλλά επειδή η διατύπωση που αποφάσισα να προσδώσω στην έκθεση αυτή, ακριβώς ε, προϋποθέτει να επικεντρωθούμε σε θέματα τα οποία είναι σημαντικά για την ΚΕΠΑ ή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει την παρουσία της, όχι μόνο προς θέματα που έχουν μια σημασία. Γιατί βεβαίω αυτά είναι εξαιρετικά πολύ άριθμα, αλλά δεν είναι εδω να συμπεριληφθούν. Αυτό είναι από του λόγου, για παράδειγμα, που η υπόδειξη του κυρίου Σιντσέβιτ να συμπεριληφθεί η Ασία δεν μπόρεσε να γίνει αποδεκτή εκ μου. Λοιπόν, επικεντρωμένη έκθεση, εστιασμένη στο διάλογο με το Συμβούλιο. Γι' αυτό σας προτείνω 14 τροπολογίες, συμβαστικές τροπολογίες. Η πρώτη αφορά τη διατλαντική ημερήσια διάταξη, η δεύτερη αφορά αρχές και αξίες τις οποίες θα πρέπει να βασίζεται η ΚΕΠΑ, η τρίτη αφορά την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας και δεν συμπέλαβε ορισμένε υποδείξει γιατί επικαλύπτονται με την έκθεση του Κάλφων Βόγκαου. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγο να πούμε στα δικά του χωράφια πέντε ε, στο, για το Κόσοβο, έξι για τη Βοσνία Ριζεγοβίνη, εφτά για την Ανατολική γειτονία, για τη γειτονία με την Ανατολική Ευρώπη ε, και σχέσεις με τις παρευξήνιες ε, χώρες Ελπίζω ο κύριος Σφάρτσαμπερκ να μας βοηθήσει να εξεύρουμε μια εύστοχη διατύπωση για τη σχέση μεταξύ Ανατολικής Γειτονίας και χωρών παρευξήνιας συνεργασίας. Μετά Ρωσία και οι σχέσεις με την Μέση Ανατολή. Δεν βλέπω εδώ το συντονιστή, ενδεχομένως θα ξεχωριστεί ψηφοφορία και μετά 12 και 13 για το καυτό θέμα του Αφγανιστάν. 14 αφορά την ε, γνωμοδότηση του, της Επιτροπής Προϋπολογισμού για το προπολογισμό της ΚΕΠΑ. Υπήρξε πολύ καλή συνεργασία, συνομίλησα με όλους τους σκιώδες συγητές από όλες τις πολιτικές ομάδες και όπως σας είπα με κάθε καλή πίστη προσπάθησα να συμπεριλάβω όλες τις παρουσιάσεις που μου υπευλήθησαν με αυτές τις δύο εξαιρέσεις όπως σας είπα Δηλαδή αν υπάρχει επικάλυψη ε, δεν συμπεριέλαβα αυτή την πρόταση. Ή εφόσον πρόκειται για θέματα τα οποία ναι μεν σημαντικά αυτά καθ' αυτά αλλά δεν βρίσκονται στο επίκεντρο της ΚΕΠΑ σήμερα ή μελλοντικά. Και αν θέλουμε να επιβάλλουμε στο Συμβούλιο, μάλλον να διαφορμόσουμε τη μέθοδο εργασίας του Συμβουλίου θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρες αναφορές στη μέθοδο εργασίας. Νομίζω ότι το Συμβούλιο ε, δέχεται αυτή την προσέγγιση όπου βαθμία ε, μέσα από την οποία βελτιώνονται βαθμία τα αποτελέσματα της εργασίας. Συνεπώς λοιπόν δεν μπορούμε να είμαστε τόσο φλίαροι. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό στα αγγλικά, λέει ο μιλητής δεν μπορούμε να καλύψουμε τα πάντα, να μιλάμε που παντός επιστητού, αν θέλετε. Σε αυτούς τους συναδέλφους, των οποίων οι, οι παρατηρήσεις συγγνώμη, δεν συμπεριλήφθησαν, ε, συμφωνώ ίσως επί της ουσίας, αλλά δεν συμφωνώ ότι ο δεδειγμένος τόπος να αναφερθούν είναι εντός αυτής της έκθεσης. Και όπως θα ε, διαπιστώσετε προσεχής έκθεση του Συμβουλίου αφορά το διάλογο αυτό ή ε, μάλλον ε, αποτελεί τμήμα αυτού του διαλόγου συμπεριλαμβάνοντας τις προτάσεις του Κοινοβουλίου. Έτσι λοιπόν θέλω να έχω μια σωστή συμπληρωματική σχέση όχι μόνο ενημερώνοντας το Συμβούλιο αλλά διαμορφώνοντας την ε, φιλοσοφία του ώστε να υπάρξει μια προστιθέμενη αξία ε, νομιμότητα στις πολιτικές αποφάσεις του Συμβουλίου. Αυτά είναι εν τα όσα ήθελα να πω εισαγωγικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και τώρα θα περάσουμε στη συζήτηση. Κυρία Κόπα. Κυρία Κοπά, ε, λέει ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σάρους Βόλσκι για την πρότασή του, διότι με τον τρόπο αυτό κατόρθωσαν καλύψει τα περισσότερα θέματα της ΚΕΠΑ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ότι κάλυψε ε, πολλά θέματα. Ευχαριστούμε και για τις ε, επικοδομητικές του προτάσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι τώρα με τους ε, συμβασμούς αυτούς έχουμε ένα πολύ πιο ισόρροπο κείμενο ανεξάρτητα με το κατά πόσο εξακολουθούν να παραμένουν διαφωνίες σε κάποια σημεία. Να επισημάνω τις βελτιώσεις η ανατολική διάσταση. Εκεί είναι σημαντικό να διευκρινιστεί η σχέση ανάμεσα σε διάφορες πολιτικές ε, όπως και να υπάρξει μια επικοδομητική συζήτηση με τη Ρωσία έτσι ώστε να εντοπιστούν ε, κάποιες ε, λήψεις ενδεχομένως που υπάρχουν στη σχέση μας με αυτή τη χώρα. Όσον αφορά την μεσογειακή πολιτική, τα πιο, τα πιο σημαντικά στοιχεία ξεκίνησαν με την ε, διαδικασία της ε, Βαρκελόνης. Αυτά παρουσιάζονται θαυμάσια στο κείμενο και αναφέρεται επίσης και ε, η προσπάθεια να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μια κοινοβουλευτική διάσταση. Σχετικά με την Αφρική, για μα είναι σημαντικό να αναφέρουμε την ανάγκη πολλών πολιτικών χωρί να εστιάσουμε την προσοχή μα μόνο σε σημαντικέ συγκρούσει, ενώ παράλληλα να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και αυτέ. Ε, για τη Λατινική Αμερική είναι σημαντικό να αναφέρουμε τι τρέχουσε διαπραγματεύσει ε, και ειδικά τώρα όπου ε, πρόκειται να υπογραφεί η πρώτη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει όμω ένα σημείο όπου δεν κατορθώσαμε να συμφωνήσουμε με τον εισηγητή. βεβαίω πρόκειται για το Ισραήλ και κυρίως για το θέμα της, Γάζα, της Γάζας. Ε, θεωρούμε ότι η αναβάθμιση των σχέσεων με το Ισραήλ δεν είναι ικανοποιητική και γι' αυτό ε, προτείνουμε συμβαστική πρόταση κατά τμήματα. Επ' αυτού διαφωνήσαμε ριζικά και ως πολιτική ομάδα αρνηθήκαμε να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση ενώ ε, υπάρχουν πολλά θέματα που είναι ανοιχτά και πρέπει να συμφωνήσουμε επ' αυτών. Θα προτιμούσαμε άλλα θέματα όπως η Βοσνία Ερσεγοβίνη ή η ανατελική διάσταση να εξεταστούν περισσότερο περισσότερο σε βάθο, παρότι βέβαια γνωρίζουμε τους ε, περιορισμούς που έχει κανείς όταν πρόκειται να παρουσιάσει μια τόσο γενική έκθεση. Σε γενικές γραμμές η δική μας ομάδα είναι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα της έκθεσης και θα θέλαμε για άλλη μια φορά να επαναλάβουμε τις ευχαριστίες μας τόσο στον κύριο Σάρου Βόλσκι όσο και στις γραμματείε των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Τελειώνω λοιπόν την παρέμβασή μου με μία μια ε, προφορική ερώτηση για τη νέα παράγραφο 22α και διαβάζω αφορά στο ε, αδιέξοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Μεσόγειο λόγω των εξελίξεων στη Γάζα και εκφράζει την ελπίδα η ευρωμεσογειακή συνεργασία να ξαναξεκινήσει στο μότερο δυνατόν και να προσφέρει τις υπηρεσίες της στον κοινό στόχο που είναι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ευχαριστώ πολύ. Λάγκεντάικ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, όπως ε, είπε και η συνάδελφός μου η Σκιώδης, η συγγήτρια, σε διάφορες άλλες περιπτώσεις, πιστεύουμε ότι η έκθεση περιλαμβάνει πολλά ικανοποιητικά στοιχεία, ε, τον αφοπλισμό, την πολυμέρεια και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πρέπει να σας πω, δεν κατανοούμε γιατί δεν υιοθετήσατε κάποιες από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν ε, που είναι καθοριστικές για τις δικές σας παραγράφους. Παράδειγμα, στην 52 την τροπολογία ισχυριζόμεθα ότι οποιαδήποτε συνεργασία στο Νότιο Κάφκασο δεν θα λειτουργήσει αν δεν λυθεί το θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Αυτή είναι μια μετριοπαθής ε, έκφραση, αλλά παρόλα αυτά δεν τη δεχτήκατε. Η 79, όπου εκφράζουμε τη λύπη μας ε, για το ότι η Κίνα σταμάτησε να συζητά με το Δαλάι Λάμα και αυτή η πολύ μετροπαθή ε, θέση και αποδεκτή του Κοινοβουλίου. Πρέπει να ομολογήσω ε, ένα, ε, μια άλλη λιγότερο επίμεχη τροπολογία, η 30, όπου διερωτώμεθα κατά πόσον πρέπει να υπάρχει αυτός ο κατάλογος τρομοκρατικών οργανώσεων. Είναι χρήσιμο, λειτουργεί. Και αυτό βασίζεται όχι τόσο στη δική μας την κρίση, αλλά σε διάφορες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που επικρίνουν κυρίως το ότι αν έχει κανείς μπει σε αυτόν τον κατάλογο είναι δύσκολο να βγει. Αυτό συζητιέται εκτός Κοινοβουλίου και είναι μια δικαιολογημένη ανησυχία. Αυτές λοιπόν είναι τροπολογίες που θα ήθελα να σας παρακαλέσω ε, να τις ξανασκεφτείτε, να δείτε αν μπορείτε να τις υιοθετήσετε. Και τέλος κύριε Πρόεδρε υπάρχει ένα λάθος νομίζω στη συμβαστική πρόταση τη δική σας την υπαριθμών 5 για το κοσυφοπέδιο. Εκεί αναφέρεται ότι η αποστολή Γιούλεξ που συζητήσαμε για αυτήν σήμερα στην έκθεσή μου για το κοσυφοπέδιο είναι ουδέτερη. Αυτό μοιάζει να είναι αλήθεια με την πρώτη ανάγνωση, αλλά δεν είναι αλήθεια. Στην έκθεση του κυρίου Μπανκιμούν ε, υπάρχει μια ε, πολύ προσεκτική διατύπωση. Λέει ότι η Ulex λειτουργεί υπό την ε, ομπρέλα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό δεν είναι σύμπτωση, δεν είναι παιχνίδι με τις λέξεις, απλά λέει ότι το καθεστώς της Ulex είναι ουδέτερο. Και νομίζω γι' αυτό στην παράγραφο υπαριθμών 5 θα ήθελα να επιδείξετε αυτό, να αφήσετε κατά μέρος αυτό που λέει ουδέτερη προς το καθεστώς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είχα δύο τροπολογίες και χαίρομαι που η τροπολογία για το Αφγανιστάν είναι πραγματικά μια πολύ καλή τροπολογία η οποία θέτει πέρασε πολλές παρανοήσεις ε, λέγοντας ότι θέλουμε, επιθυμούμε τις συζητήσεις με όλες τις ε, πολιτικές ε, ομάδες στο Αφγανιστάν εφόσον ε, αποκηρύξουν τις τρομοκρατικές ενέργειες. Τώρα όσον αφορά την παράγραφο 72 για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ. Καταρχήν όσον αφορά την υποστήριξη της των δημοκρατικών διαδικασιών και ιδιαίτερα, κατά ο λόγο, ε, σε υποστήριξη της αποστολής ε, EULEX, ε, της οποίας θετία παρατείνεται. Θα ήθελα να συστήσετε στα μέλη να υποστηρίξουν αυτή την τροπολογία υπαριθμών 72. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω για την τροπολογία υπαριθμών 67 και τις τροπολογίες 20 και 10 και εκτό. Υπήρχαν, υπήρξαν πολλές ε, δύσκολες διαπραγματεύσεις όσον αφορά την κατάσταση στη Γάζα και στο Ισραήλ, ε, μια συζήτηση για το τι θα γίνει πριν από τα Χριστούγεννα. Είναι πολύ δύσκολη η επίτευξη μια συνένεση εκ μέρους όλων των πολιτικών ομάδων. Ε, το θέμα του Αμπού Γκράιπ δεν πρέπει να αναφερθεί σε άμεση σύνδεση με τη Γάζα. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ανθρωπιστική κατάσταση και στην άμεση ανασυγκρότηση. Ε, το Συμβούλιο θα πρέπει να σχολιάσει για το Αμπού Γκράιπ. Αυτή ήταν μια συνένεση μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων. Συνεπώς λοιπόν θα ήθελα να επαναθεωρήσετε το 20 α ε, well... της συμβαστικής πρότασης 10. Ε, αν κατάλαβα καλά, τα όσα συμφωνήσαμε για, στο συμβασμό για τη Γάζα ήταν... Ε, εγώ είχα μια άλλη άποψη. Αποφασίσαμε να βάλουμε στις αιτιολογικές σκέψεις ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επιθυμεί μια αναβάθμιση της σχέσης. Δηλαδή, αφαιρέσαμε το κείμενο αυτό από το τέλος του ψηφίσματος και το βάλαμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Δεν συμφωνώ λοιπόν με το αίτημα της κυρίας Ιμπάσκοβα, ενώ συμφωνώ με τα όσα λέει το κείμενο. Εγώ θα προτιμούσα να μείνουμε στη θέση στην οποία συμφωνήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, επιφυλάσσεται της ε, συγκατάθεσή του. Ε, επιφυλασσόμενο κατά πόσο η κατάσταση θα αλλάξει όχι. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση και η προσέγγιση της δικής μου ομάδας σχέση με το θέμα αυτό. Ωραία, θα δώσω πάλι το λόγο στην κυρία Ιμπάσκοβα και στη συνέχεια στον εισηγητή, τον κύριο Σάρος Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε το λόγο εμείς στις διαπραγματεύσεις ε, περάσαμε στη ε, θέση της δήλωσης ε, χωρίς να τίθενται κάποιοι όροι. Αυτό αποδέχτηκε από όλες τις πολιτικές ομάδες. Ήταν η γραμμή την οποία διαπραγματεύτηκαν και στην οποία συνήνεσαν όλες οι πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Σαρισβόλσκι έχει τώρα το λόγο για τις καταληκτικές ε, παρατηρήσεις. Ωραία. Ε, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε συμπληρωματικοί με τις πιο λεπτομερικές εκθέσεις της ΑΦΕΤ. Δεν είναι δυνατόν να ικανοποιήσουμε όλους χάνοντας τελικά τον στόχο μας ναι μεν ε, συμφωνώ με πολλές απόψεις, αλλά αν συγκεράσουμε όλες τις απόψεις τελικά θα πάψει να είναι εύληπτο το κείμενο και θα χάσουμε το στόχο. Γι' αυτό εφαρμόζω μία αυστηρή λογοκρισία. Αλλιώς το κάθε άρθρο θα γίνει ένα ψήφισμα. Πρόκειται για ένα για μια έκθεση κατά δεύτερο λόγο η οποία ε, θα διατηρήσει ένα επίκαιρο χαρακτήρα για ορισμένους ε, μήνες. Εάν συμβεί κάτι την επόμενη Δευτέρα, ε, δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτά τα θέματα και αυτό το σκοπό έχουμε άλλωστε τα κατεπήγοντα. Τώρα, αν επανέλθουμε στις παρατηρήσεις των συναδέλφων, θα ήθελα να πω το εξή. Κυρία Κοπά, όσον αφορά την ανατολική διάσταση και τη Ρωσία, η ανατολική, για την ανατολική διάσταση, διάσταση γειτονία με τις ανατολικές χώρες, είχαμε μία συζήτηση και θα υπάρξει μια, ένα σχετικό ψήφισμα. Γι' αυτό δεν ήθελα να επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Στην ε, Μεσογειακή Ένωση, ε, για τη Μεσογειακή Ένωση νομίζω ότι είπατε για το συμβιβασμό 11 Euromed είστε ικανοποιημένοι. Για την Αφρική και τη Λατινική Αμερική δεν υπάρχει συμφωνία για τη Γάζα. Και έχοντα ακούσει τα όσα είπε η κυρία Ιμπάσκοβα, θα πρότεινα να αποσύρουμε όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί ε, ορισμένοι δεν επιθυμούν να συμπεριληφθεί. Ορισμένοι δεν θέλουν να, να συμπεριληφθεί. Υπάρχει διαφωνία λοιπόν, άρα καλύτερα να αποσυρθεί. Το θέμα είναι κατά πόσο τα διέξοδα στην Ευρωμεσογειακή Ένωση οφείλονται στη Γάζα. Γιατί εκεί η σχέση μεταξύ των δύο δεν είναι τόσο απλή. Εάν επιμείνετε μπορούμε να ζητήσουμε σχετικά νομίζω ότι όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται σε ένα εστιασμένο ευρωμασογικό ψήφισμα. Γι' αυτό ας μην κάνουμε τέτοιου είδους αξιολογήσεις συνθετικής φύσεως όπου θα δώσουν λαβή σε περισσότερες παρανοήσεις. Τώρα, στα όσα είπε ο κύριος ε, Λαγκεντάκ, έχετε δίκιο τον Αγκόρνο Καραμπάχμεν, αλλά δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε κάθε σύγκρουση που έχει παγώσει, γιατί αλλιώς θα πρέπει να έχουμε ακόμα 10-15 παραγράφους για την Κίνα. Ε, τις ανησυχίες για το Θιβέτ, δεν έχει γίνει τίποτα και εμείς ε, ε, απήχαμε παντελώς και ακριβώς γι' αυτό δεν το αναφέρω. Ε, λοιπόν, συμμερίζομαι την διάγνωση που κάνατε αλλά μοιάζει να υπάρχει μια πλήρη ανικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Κίνα και, τα ανθρώπινα, και τη θέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί. Τώρα, στο 30... Δεν ξέρω, σε σχέση με τη χρησιμότητα των δημοκρατικών καταλόγων. Νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο θέμα και ίσως θα έπρεπε να παρεμφευθεί στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μπούμε σε τόσο επικίνδυνα νερά. Στην EULEX ε, ε, ε, συμφωνώ. Τώρα, για το 72, για το Ιράκ θα το εξετάσουμε. Κυρία Ιμπάσκοβα, έφυγε η κυρία Ιμπάσκοβα, αλλά θα αποσύρουμε το upgrade. εάν δεν θέλουμε να το αναφέρουμε. Είναι γνωστό σε όλους ότι αυτό το κοινοβούλιο δεν έδωσε την συγκατάθεσή του στο upgrade. Ας το αφήσουμε λοιπόν, ας το αφαιρέσουμε. Αυτά είναι όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Και αν αυτό είναι όλο, τότε να σας ότι θα ψηφίσουμε αύριο. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα. Ε, βλέπω να είναι εδώ κοντά μας ο εισηγητής μας, ο κύριος ε, Φον Βόγκα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, καταρτίζοντας αυτή την έκθεση για την στρατηγική ασφάλεια, αντιμετωπίσαμε τη δυσκολία το Συμβούλιο να καθορίσει και να ολοκληρώσει τη στρατηγική του μόλις στο τέλος του προηγούμενου έτους. Άρα δηλαδή εμείς είμαστε αναγκασμένοι να εργαστούμε πάνω σε κάποιες εικασίες για αλλαγές που θα έκανε το Συμβούλιο. Θέλω όμως να σας πω ότι είμαστε ευγνώμονες ε, στο Συμβούλιο και τους εκπροσώπους του. Εργαστήκαμε πολύ στενά, ανταλλάξαμε πληροφορίες, έτσι λοιπόν ε, μπορούσα να προβλέψω κατά κάποιον τρόπο ε, πώς ακριβώς θα διαμορφωνόταν η πρόταση της Προεδρίας. Μία δεύτερη δυσκολία είναι η εξή και τώρα φτάνω στις ε, συμβαστικές ε, προτάσεις ε, στο άρθρο 9 γίνεται λόγος για τις φιλοδοξίες της Γαλλικής Προεδρίας επειδή μεταξύ έχει τελειώσει η Γαλλική Προεδρία Πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τη λέξη εδώ ambitions και να προσθέσουμε τη λέξη initiatives, ε, πρωτοβουλίε στα αγγλικά. Ε, θα μου επιτρέψετε με λίγα λόγια να σας ε, παρουσιάσω τα βασικά σημεία της έκθεσής μου. Γιατί έχει κατατεθεί μια μεγάλη σειρά τροπολογιών που εγώ τις, έχουμε τροπολογίες που τις δέχομαι. Άλλες που έχω καταθέσει και εγώ. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αναφέρω την κεντρική ιδέα της έκθεσης. Αφενός το γεγονός ότι η στρατηγική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, επανεξετάστηκε. Αυτό το βρίσκω σωστό. Ε, πρόκειται για προσαρμογή σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχουν τροποποιηθεί. Νομίζω ότι στο μέλλον ε, θα πρέπει αυτό αναφέρεται και σε ένα άρθρο της πρότασης. Θα πρέπει λοιπόν στο μέλλον κάθε ε, αμερικανική κυβέρνηση όταν αναλαμβάνει να παρουσιάζει μια στρατηγική ε, ασφάλειας και μετά κάθε χρόνο να ε, μπορούμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η στρατηγική αυτή έτσι ώστε ανά πέντε χρόνια θα έχουμε και μια στρατηγική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε μια γενική εικόνα του τι ακριβώς συνέβη. Κατόπιν, Όσον αφορά ε, το σχέδιο που σας έχει κατατεθεί, έχουμε τη δική μας την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας που εστιάζεται κυρίως στην πρόληψη, την διαχείριση κρίσεων και τη συνεργασία του στρατιωτικού με τον πολιτικό τομέα. Οφείλουμε να δράξουμε την ευκαιρία ε, για να ε, επανεπεξεργαστεί και το ΝΑΤΟ τις δικές του απόψεις περί στρατηγικής ασφάλειας. Αυτά θα τα πει μάλλον στο Στρασβούργο και στο ΚΕΛ και από ό,τι φαίνεται αυτή η στρατηγική ασφαλείας του ΝΑΤΟ θα ισχύει για ένα χρόνο. Αυτή η παράλληλη συζήτηση θα πρέπει να αποτελεί το έναυσμα έτσι ώστε να ε, προσπαθήσουμε να φέρουμε πιο κοντά το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική μου έκθεση εστιάζει στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί νομίζω ότι στην Ένωση έχουμε αξίες που πρέπει να υπερασπιστούμε, αλλά και συμφέροντα τα συμφέροντα της Ένωσης και των πολιτών της. Όσον αφορά τα συμφέροντα πρόκειται για την εξασφάλιση των εξωτερικών συνόρων, ε, της, ε, της υποδομής, ε, προστασία από τρομοκρατία, από όπλα μαζικής καταστροφής, ενέργεια, κλιματική αλλαγή. Αυτά είναι λέξεις κλειδί που τις βρίσκεται τις λέξεις αυτές στην έκθεση. Και ένα κεφάλαιο για τη Ρωσία σε σχέση με τη Γεωργία. Η έκθεση θεωρεί ότι η αντίδραση της Ρωσίας ήταν δυσανάλογη. Βεβαίως και από την πλευρά της Γεωργίας ε, διεπράχθησαν λάθη. Στην πρόταση της έκθεσης αναφέρεται ότι ε, το αίτημα του Τόμας Ήρβης η στρατηγική του ΝΑΤΟ για τις ε, χώρες, ε, για την ε, άμυνα των χωρών της να συγκεκριμενοποιηθεί. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα στην έκθεση. Γνωρίζω ότι το θέμα αυτό θα παραμείνει επίμαχο. Άλλα θέματα είναι ενέργεια και απόκρουση πυράβλων. Εδώ επικρατούν διαφορετικές απόψεις στην Επιτροπή μας. Υπάρχει άποψη ότι η απόκρουση πυράβλων δεν θα συνεχιστεί από τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση. Εγώ βέβαια δεν είμαι πεπισμένος γι' αυτό ε, λόγω όλων αυτών που ακούσαμε και από τον Υπουργό Εξωτερικών κύριο Σβάτσενμπεργκ. Κατόπιν στην έκθεση ακούτε ή βλέπετε κάποιες ε, ικανότητες ε, που είναι απαραίτητες. Νομίζω εδώ η τροπολογία του συναδέλφου κυρίου Κούνε, η τροπολογια του αδελφου κυριου κουνε η υπαριθμον 62 είναι πολύ σημαντική, γιατί ε, κατ' ουσίαν η τροπολογία αυτή υιοθετεί ακριβώς εκείνα ε, τα οποία αποφάσισε το Συμβούλιο κατά ε, τις ε, τελευταίες εβδομάδες του περασμένου έτους. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να υπάρχουν μόνο 60 μέρες στη διάθεσή μας, αλλά να είναι και πολύ συγκεκριμένο το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω από όλα αυτά ε, μπορεί κανείς να εξάγει το ότι πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά, να βελτιωθούν οι ικανότητες ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρχουν ηγετικές δομές, επιχειρήσεις, βελτίωση της στρατιωτικής με την πολιτική συνεργασία ε, να, υπάρχουν, ε, ε, να υπάρχει εδώ η έδρα στις Αυτά είναι κάποια αιτήματα που αναφέρω έτσι ενδεικτικά. Επίσης γίνεται αναφορά και στους εξοπλισμούς. Αυτό έχει γίνει και σε παλαιότερες εκθέσεις. Και τέλος υιοθετώ μία έννοια την οποία κατά κύριο λόγο παρουσίασε ο κύριος Πέτερινγκ Synchronized Armed Forces Europe. Αυτό που είναι καινούριο είναι ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε την κοινωνική κατάσταση των ε, στρατιωτών που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. παραδείγματος χάρη είναι εξασφαλισμένοι. Οποτεδήποτε ε, υπάρχουν επιχειρήσεις όπου πεθαίνουν οι ε, στρατιώτες αυτοί διαπιστώνουμε ότι στις περιπτώσεις αυτές ε, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και που ακόμα υπολείπονται. Και τέλος υπάρχει και ένα δικό μας αίτημα που είναι η στρατηγική ασφάλειας να συγκεκριμενοποιηθεί κατά την επόμενη θητεία μέσα από λευκή βίβλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ως πρότυπο μπορούμε να πάρουμε την γαλλική λευκή βίβλο που περιλαμβάνει και ένα μεγάλο ευρωπαϊκό κομμάτι. Η Γαλλία ενδιαφέρεται για όλα αυτά. Ε, έγιναν πολλές συζητήσεις ε, στη Γαλλία, πάρα πολλές ακροάσεις που ήταν και ανοιχτές για το κοινό. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι εκείνα, ότι όλα αυτά μπορούμε να τα υιοθετήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί κατ' ουσίαν αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια ανοιχτή συζήτηση για την πολιτική άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά δεν θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα και κλεισμένων των θυρών, αλλά ε, θα πρέπει να υπάρχει μια αρκετά εκτεταμένη συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φων Βόγκαου, ε, σκιώδης ε, εισηγητής ε, εκ μέρους των σοσιαλιστών. Είναι ο κύριος Χέλμουντ Κούνε και έχει το λόγο. Δεν θα με ακρηγορήσω. Έχω να σας πω τα εξής. Πρώτα πρώτα κάτι διαδικαστικό για να μην δημιουργούμε σφαλμένες εντυπώσεις αποσύρω την τροπολογία παριθμών 1 γιατί δεν διαπιστώνω να υπάρχει πολιτική βούληση ούτω ώστε να αποφύγουμε επικαλύψεις με προηγούμενα ψηφίσματα επομένω, αύριο ε, θα ψηφίσουμε το ίδιο πράγμα, το ίδιο αίτημα για τρίτη φορά. Ε, ε, το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχει αυξημένο ειδικό τώρα, κάτι άλλο τώρα, ε, κάποιο είδους άκομψες εκφράσεις, άτσαλες, έχουμε αυτό το cyber warfare κυβέρνο πόλεμος λέγαμε κυβέρνο επιθέσεις στο παρελθόν Προσέξτε γιατί με το χρησιμοποιούμε αυτό θα υπάρχουν συγκεκριμένε ε, συνέπειε. Δηλαδή, θα, ε, εάν λέμε ότι αυτό είναι πράξη πολεμική, πράξη πολέμου, τότε θα πρέπει ε, και η απόκριση να είναι επίσης πολεμική πράξη. Άμα τα θέλουμε αυτά τα πράγματα τότε καλή μας τύχη. Μας ακούτε? Όχι. Off the Baltic states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 Πάλι εδώ πέρα έχουμε αδόκιμη έκφραση. Αν θέλουμε εδώ να θέλουμε να είμαστε έτσι απλά η φωνή του ΝΑΤΟ και στη συνέχεια θέλουμε ε, να υπάρχει κάποιο είδους προγραμματισμός της άμυνας αυτό σημαίνει ότι υπάρχει υπαρκτή απειλή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το μάθαμε δεκαετία του 70 και 80. Άμα το κάνει κανείς αυτό, τότε έχουμε αυτή τη σπήρα, αυτό τον φαύλο κύκλο της ρητορική και της διατύπωσης απειλών, διότι ο κύριος Νταφ και εγώ ε, έχουμε μια τροπολογία προφορική που θα σας την διαβάσω. Α, είναι υπέροχη τεχνολογία που μας περιβάλλει. Λαμβάνει υπόψη ε, ότι επιβεβαιώνει το ΝΑΤΟ και τα κράτη-μέλη το ότι συνεχίζει να ισχύει το ότι ε, κατησχεί το άρθρο 5 της συνθήκης του Βαταντικού Συμφώνου. Δεν ξέρω, είσαστε ικανοποιημένοι γιατί χρειάζεται όντως να συμμορφωθεί κανείς προς το 5 Συμφωνούμε, αλλά όχι παραπέρα. Εγώ θεωρώ ότι ο πρόεδρος Ομπάμα θα χρειαστεί τα χρήματα για άλλους σκοπούς και όχι για τέτοιου είδους τρίτης, τέταρτης κατηγορίας προγράμματα της κυβέρνησης Μπούς. Ε, ενδεχομένως βέβαια τα έχει υπολογίσει κατά άλλο τρόπο όσον αφορά Ιράν και Ρωσία. Καλά, δεν θέλω τώρα να κάνω τέτοιου είδου μαντεψίες. Ε, Αυτό αφορά και το ε, αντιπυραυλική ασπίδα. Εμείς θέλουμε να απαλληφθεί αυτή η παράγραφος, κάντε εσείς ό,τι θέλετε. Όλοι εκείνοι οι οποίοι με επιφύλαξη είναι υπέρ αυτή τη υπόθεση, Για πετε μου, όντω θεωρείτε ότι τη σήμερα μέρα μία μέρα μετά από την ορκομοσία του κυρίου Ομπάμα, όντω πιστεύετε ότι ο κύριος Ομπάμα υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει αυτή την υπόθεση όχι για μην κάνετε τον ήρωα για μην κάνετε τους τελευταίους σουλιώτες στο, στο κούγκι για τους Και εγώ, πρόεδρε, θα ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Καρλφόν Βογκάου διότι ε, έδωσε δυναμισμό στο σχέδιο κειμένου τώρα δε είναι ξεκάθαρο το ότι απέτυχαν τα κράτη-μέλη αλλά και το Συμβούλιο να ε, μπορέσουν να διατυπώσουν κάπως αυτές τις φιλοδοξίες για την ασφάλεια και τη στατική της που ξεκίνησαν το 2003 ένα γιατί δεν είχαμε καθόλου πρόοδο. Τόσο το μάλλον αφού παγκοσμίως απαιτείται περισσότερη ασφάλεια και λέμε τώρα για το τι έγινε τους τελευταίους μήνες. Ο δε εισηγητής κατάφερε όλα αυτά να τα εντάξει στις εύστοχες τροπολογίες του. Στην δε υπαριθμών 2 ε, θα πρέπει να συγχαρούμε την Γαλλική Προεδρία για την ΚΕΠΑ και η δε ιστορία και ιστορική θα μπορέσουν να δουν βέβαια με κριτικό μάτι τα υπέρ και τα κατά τη Γαλλικής Προεδρίας όσον αφορά την ε, κοινή εξωτερική πολιτική. Όμως έπρεπε να υπερκυράζει κάποια, κάποια εμπόδια η Γαλλική Προεδρία και βέβαια οι άλλοι πώ να το ε, καταφέρουν αλλά λέει ιστορία γιατί ήταν ε, κρύοι και φλεγματικοί και αγοκολώνες, δεν ανταποκρίνονται οι Βρετανοί όσον αφορά όλα αυτά τα υπομορφή πρόκλησης που έβαζαν στο τραπέζι οι Γάλλοι. Ελπίζω ότι πιο θετικά και πιο γρήγορα θα τα δει η κυβέρνηση της χώρας μου όσον αφορά την ε, ε στατική ασφάλεια Περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Για τις βαλτικές χώρες Συμφωνώ 100% με τον κύριο Κούνε. Μας εξήγησε και πώς έχει η τροπολογία του η οποία θεωρώ ότι είναι επαρκέστατη για όλους μας. Δεν θα πρέπει το Κρεμλίνο να θεωρήσει ότι ε, πρόκειται περί προκλήσεως. Αυτά όσον αφορά την παράγραφο 30 Σήμερα να σας πω την αλήθεια. Δεν επίστην από τον κύριο Σβάρτζεμπεργκερ όσον αφορά το αντιπροβλητικό σύστημα που υποτίθεται θα τοποθετηθεί εις Πολωνία και Τσεχία. Δεν θεωρώ ότι έγινε με το timing αυτή η ενέργεια, ότι υπήρχε κατάλληλη πολιτική ευαισθησία ή ότι δεν είναι πάρα πολύ θετικό το ότι προχώρησαν χωρίς να υπάρξει κάποιο είδους ε, ε, διαβούλευση με τους Ευρωπαίους εταίρους τους πάντως μας το είπε ο πρόεδρος Κούνε ότι ο πρόεδρος Ομπάμα κάνοντας την ε, παραθενική του ομιλία ακούσαμε πως τα είπε και θα ήταν λάθος να κάνει κάποια κίνηση που πρέπει να σκεφτεί καλά το κοινοβούλιο. Γιατί πρόκειται για αναγκαία αντιδρασή μας η οποία και θα ολοκληρωθεί εν ευθέτω χρόνο. όταν το τοπίο ξεκαθαρίσει καλύτερα και περισσότερο στο μέλλον. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος και το λόγο στον κύριο Λάχεντάικ για τους πρασίνους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά από τα όσα είπαμε την Αγγέλη Γαμπίερ τη συνάδελφο, δεν θα εκπλήξω και τον εισηγητή για το ότι δεν είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι για να το πω έτσι διπλωματικά για την έκθεση μια που θεωρούμε ότι είναι παράδοξο πάλι το λέω διπλωματικά όσον αφορά το πού ξεχωρίζει η Επιτροπή Ασφάλειας η, η, η Στατική Ασφάλειας όπως λέει ο κύριος Βατάνεν λέει ο κ. Βατάνεν ότι έχει μοναδικές ικανότητες όσον αφορά την αποτροπή συγκρούσεων και επίλυση των κρίσεων και όσον αφορά μηχανισμούς για τις ανθρωπιστικές κρίσεις εδώ, σε αυτή την έκθεση θα έπρεπε να μπουν τέτοιοι χαρακτηρισμοί, όχι στην έκθεση ΝΑΤΟ Βατάνιν, αλλά στην έκθεση που τώρα συζητούμε για στατική ασφαλεία. Γιατί ο εισηγητή δεν θέλει εδώ να ασχοληθεί με κάποιε έννοιε που δεν είναι και τόσο προοδευτικέ ή αριστερέ, α πούμε. Το ότι ε, όπως είπε και ο ΙΕ θα πρέπει να υπάρχει μέσα στην ασφάλεια και ενίδες προστασίας 55 έως 67 ε, σε αυτές τις διατάξεις δεν καταλαβαίνω γιατί εκεί, εκεί δεν περιλαμβάνει κάποια άλλα στοιχεία για την κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική το, το ίδιο σκεφτόμαστε και για το ότι αρνείται ο συγητής ακόμα και να μνημονεύσει τη συνθήκη για την μη διάδοση των πυρηνικών και για συγκεκριμένα το θέμα του αφοπλισμού γιατί εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακόμα και στη ΣΥΠΑ γίνεται κουβέντα για αυτό το πράγμα για την αφοπλισμό στα πλαίσια της συνθήκης αυτής άρα αυτή η συνθήκη θα έπρεπε τουλάχιστον να μνημονεύεται και δεν ξέρω γιατί δεν το έχει κάνει Γι' αυτό και θεωρώ ότι εάν δεν αλλάξει τη θέση του εισηγητής εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής ε, μας πέστη την προσοχή σε ένα βασικό πρόβλημα το οποίο νομίζω συμμερίζονται όλες οι πολιτικές ομάδες, δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας, η, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφαλείας ε, έγινε σε μια στιγμή που το, η έκθεση αυτή βρισκόταν υπό εξέλιξη. Και ε, συνεπώς η παρούσα κατάσταση των πραγμάτων δεν μπορεί να αντικατοπτριστεί επαρκώς αυτή την έκθεση. Γι' αυτό θα ήθελα να το πούμε αυτό και ρητά στην έκθεση. Ενδιαφέρον το συνάδελφος Κούνα στην τροπολογία του υπαριθμών 63 στο πρώτο ε, τμήμα, στο προσινό τμήμα το περιγράφει νομίζω σωστά. Το υπόλοιπο δεν το υποστηρίζουμε πολιτικά. Δηλαδή λέει ότι το δεν υπήρξε διαβούλευση με το κοινοβούλιο. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι γεγονός και θα ήταν η επιθυμία μου να συμπεριληφθεί αυτή η φράση. Ενδιαφέρον βρίσκω κύριε Φων Βογκάου το γεγονός ότι στην τροπολογία υπαριθμών 20 της συναδέλφου Αγγέλικα το πρώτο τμήμα ε, στηρίζεται το πρώτο τμήμα ε, της ε, έκθεσης της κοινοβουλευτικής της έκθεσης της για την ευθύνη του Κοινοβουλίου αλλά όχι στη συνέχεια και πραγματικά αυτό με σοκάρισε λίγο με σοκάρισε το ότι δεν τονίζεται τη σημασία του διεθνούς δικαίου ελπίζω ότι αύριο θα καταφέρουμε να συμπεριληφθεί το θέμα του διεθνούς ε, δικαίου εδώ σε συνεργασία με τις άλλες πολιτικές ομάδες, τουλάχιστον ε, με τους ε, σοσιαλιστές και τους φιλελευθέρους. Όσον αφορά το κοινοβουλευτικό έλεγχο, είπα ότι αυτό είναι ένα σημείο όπου συμφωνεί όλη η Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας. Σας στηρίζουμε απολύτως ως προς το σημείο αυτό στην έκθεση. Ενδιαφέρουσα βρίσκω την άποψή σας για τη γεωργία, την οποία συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση. Δηλαδή λέτε ότι η Ρωσία θα πρέπει να αντιδράσει στην αντιπαράθεση αυτή. Διερτώ με πώς μπορεί να αντιδράσει σε μια αντιπαράθεση αν δεν αναφέρει ε, μεταξύ ποιον έχει συμβεί αυτή η αντιπαράθεση. Ε, δεν ξέρω ε, αν θα πρέπει να πει κανείς ποιος ξεκίνησε αυτόν τον ε, πόλεμο. Όσον αφορά το αντιπερευλικό σύστημα, ε, συμμερίζομαι τις απόψεις του κυρίου Κούνα και του κυρίου Ντάφ και ελπίζω να περάσει αυτή και ελπίζω και να αφαιρεθεί ε, αύριο βάσει της ψηφοφορίας. Τώρα η Σύμβαση για τον Εφοπλισμό θεωρώ ότι και αυτή είναι ε, σημαντική πτυχή που δεν θα πρέπει να μην συμπεριληφθεί. Ε, εν γέννη θα μπορούσαμε να πούμε ότι η έκθεση ε, πηγαίνει στην εσφαλμένη κατεύθυνση. Είναι υπέρ πολιτικής και στρατηγικής συνεργασίας. Ε, η, σχέση με τον ΝΑΤΟ έτσι όπως περιγράφεται εδώ είναι προβληματική και ε, συνολικά χαιρετίζει την διεύρυνση της στρατηγικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχει μια τροπολογία εκ μέρους μας που λέει ότι δεν επιθυμούμε αυτή την διεύρυνση στρατηγικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιθυμούμε να είναι πολιτικός και ο στρατηγικός παράγων Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο εμείς Στην ε, ψηφοφορία θα θέσουμε κάποια σημεία ε, και πραγματικά περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία τα αποτελέσματα της ε, ψηφοφορίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κατ' να συγχαρώ τον κύριο Φων Βογκάου για την εργασία του σε αυτή την έκθεση. Νομίζω ότι τόσο η έκθεση όσο και οι προταθέντες συμβιβασμοί είναι ε, πραγματικά ένα πολύ καλό σετ συστάσεων και μια καλή βάση ανάλυσης για την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Ωστόσο υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία θα εμπλουτίσουν πιστεύω την έκθεση. Πιστεύω καταρχήν ότι θα πρέπει να σημειώσουμε δύο πράγματα εμφατικά στην έκθεση. Ότι οι συνδυασμένες επιπτώσεις της αύξησης του κόστους της άμυνας, του εξοπλισμού άμυνας. Αύξηση με την οποία είμαστε αντιμέτωποι όλοι μας. Καθώς και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες μέλη σχετικά θα πρέπει να ξεπεραστούν ή να αντιμετωπιστούν. Νομίζω ότι υπάρχει τροπολογία υπαριθμών 16 που αναφέρεται στο ότι χώρε μέλη θα πρέπει να συνδυάσουν τους πόρους και τις δυνατότητες τους ούτω ώστε να αντισταθμίσουν αυτά τα αρνητικά στοιχεία, ιδιαίτερο σε εποχέ κρίσης όπω είναι η τωρινή. Δεύτερον, νομίζω ότι είναι πολύ καλό για αυτή την έκθεση να σημειώσουμε μια σημαντική πρόσφατη εξέλιξη το Νοέμβριο η απόφαση, να συσταθεί ένας ευρωπαϊκός αεροπορικός στόλος. Νομίζουμε ότι είναι ζωτική σημασία για το Κοινοβούλιο να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία. 15 υπουργοί από 15 χώρες είναι υπέρ αυτής της πρωτοβουλίας. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω μία ερώτηση, ένα ζήτημα τεχνικής φύσεως που αφορά την παράγραφο 13 όπου ο συγητής αναφέρεται στην κρίση στη Γεωργία η οποία βήθησε τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ρωσία σε μία κρίση. Δεν ξέρω, έχετε, σημειώσατε ε, τα σημάδια αυτής της κρίσης διαπιστώσατε να υπάρχει κάποια κατάρρευση των σχέσεών μας με τη Ρωσία ή έστω κάποια κρίση. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο ακριβείς με όρους πραγματικότητας. Δεν νομίζω ότι κανείς παρατήρησε μια κρίση λόγω της γεωργίας. Ε, η κρίση θα μπορούσε να υπάρξει λόγω του φυσικού αερίου αλλά όχι λόγω της γεωργίας. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να αναφέρονται τέτοιες φράσεις που δεν αντανακλούν την πραγματικότητα. Ποτέ δεν υπήρξε κρίση με τη Ρωσία λόγω αυτής της σύραξης παρόλο που ορισμένοι πιστεύουν ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να έχει πιο στεναρό ρόλο έναντι αυτής της κρίσης. Ευχαριστούμε. Κυρία Κοπά. Ε, Ευχαριστώ και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Ευχαριστώ για την έκθεσή του και για την προστασία που κατέβαλε σε σχέση με τις τροπολογίες και ευχαριστώ επίσης και με τον κύριο Κούνε τον σκιώδη συγητή. Όμως να σταθώ στα εξή ζητήματα. Κανείς δεν μπορεί να ανηθεί ότι χρειαζόμαστε μια σφριγγυλή εξωτερική πολιτική για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις και επομένως πρέπει να συνεργαστούμε με τους άλλους παίκτες της διεθνούς κοινή ή στα πλαίσια των όσων ορίζει ο χάρτης των Εθνών και για άλλη μια φορά θα πρέπει να πούμε ότι μένουμε πιστοί στην πολυμερή ε, άποψη των πραγμάτων και ότι θέλουμε να υπάρξει αναθεώρηση του χαρτών του ΟΗΕ ούτως ώστε ε, έτσι να υπάρχει πιο σωστή διαχείριση των κρίσεων. Επίσης θα ήθελα να υποβάλω μια προφορική τροπολογία αφορά τον οργανισμό ασφάλειας ε, γιατί θα πρέπει να σταθούμε ε, στον ρόλο αυτού του διεθνούς οργανισμού όσον αφορά τον εκδημοκρατισμό και την ε, θεωρεί ότι θα πρέπει τα κράτη με την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλουν όσον αφορά τη βελτίωση του στήματος του Οργανισμού Ασφάλειας για την Ευρώπη και επίσης ότι πρόκειται για πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, επίσης ε, πρόκειται για κάτι πάρα πολύ βασικό ε, μια που έτσι θα υπάρξει η επίλυση κάποιων καταστάσεων σύγκρουσης θα έχουμε καλύτερο συντονισμό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΑΣΕ και επίσης έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε την κατάλληλη πρικοδότηση αλλά και το νομικό υπόδοση, την νομική προσωπικότητα για να μπορεί αυτός ο οργανισμός να φέρει πέρα στη σημαντική του αποστολή. Thank you, uh, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να συγχαρώ τον Καλφον Βόγκα για το έργο το οποίο επετέλεσε αλλά επίσης και για την τόσο θετική του στάση όσον αφορά τις τροπολογίες τις οποίες του παρουσιάσαμε για την εκθεσή του. Χωρίς να κολλήσει εγώ, έχω να σας πω ότι έχω την τροπολογία υπαριθμών 2. Αυτή αφορά την παράγραφο 9. Και θα έλεγα ότι θα ήταν καλύτερα εάν εκεί που λέει απειλές κυβέρνων επιθέσεων αυτό να το διατυπώνω με διαφορετικό τρόπο. Καταλαβαίνω και συμφωνώ ότι στον κυβερνοχώρο ε, υπάρχει ανάγκη ασφάλειας και προστασίας αλλά μπας και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετική ε, διατύπωση ούτως ώστε να υπάρχουν ε, κάποια μέτρα για την προστασία ε, γιατί εδώ έχουμε διάφορα ζητήματα θέματα υπηρεσιών πληροφοριών, αντικατασκοπίας, συλλογή πληροφοριών κλπ. κλπ. Κάτι άλλο τώρα όσον αφορά την τροπολογία υπαριθμών 62 του κυρίου Κούνε συμφωνώ με την τροπολογία διότι πρόκειται ε, για πάρα πολύ σημαντική τροπολογία και εδώ συνδέεται αυτό το ζήτημα με κάτι άλλο το οποίο αφορά την έκθεση πρόκειται για το ότι θα πρέπει να έχουμε τα μέτρα τα μέσα τα οποία χρειάζονται τόσο ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται αλλά υπάρχει ένα τρίτο κεφάλαιο πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο αφορεί τον εξορθολογισμό των προϋπολογισμών ούτως ώστε να μπορέσουμε να ενατενίζουμε το μέλλον πιο λογικά πιο βιώσιμα όσον αφορά τον προϋπολογισμό ή τους προϋπολογισμούς για την άμυνα. Κάτι τελευταίο το οποίο αφορά την κοινοβουλευτική διάσταση κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει όλους εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και γι' αυτό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που συνεχίζουμε εδώ να ασχολούμεθα με την κοινοβουλευτική διάσταση και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο για τα πάντα όλα όσα έχουν σχέση με την άμυνα. Τέλο δε, το κεφάλαιο για τις είπα. Βεβαίω και είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και γι' αυτό θέλω ο Καρλ να κρατήσει αυτό το θέμα ανοιχτό διότι έχουμε τώρα καινούργια Αμερικανική κυβέρνηση. Αν τώρα πήγαινε στην τηλεόραση, ανοίξτε και θα δείτε ότι έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία ανέλυψη των καθηκόντων του Προέδρου. Μάλλον αρχίζει τώρα που μιλάμε. Όμω, παραδείγματο αυτό το οποίο χρειάζεται ή να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες και ε, ποια είναι η λογική προσέγγιση ε, θεωρούμε ότι θα έχει ο κύριος Ομπάμα και η δική του για μια σειρά θεμάτων. Φυσικά και υπάρχουν κάποια θέματα, κάποιες ας προκαταλήψεις ε, στην πολιτική που ασκεί, είπα πούμε για, τις, για τα όπλα. Ελπίζουμε θα υπάρχει καινούργια προσέγγιση, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρί να μπορούμε να ξέρουμε το περιεχόμενο και είναι επίση πάρα πολύ νωρί για να ξέρουμε ε, τα, τα, τα, υπόλοιπε μεταβλητέ, δηλαδή τη στάση ας πούμε του Κογκρέσου. Τι θα μπορούν για τις προτάσεις που θα κατεβάσει ο κύριος Ομπάμα από αύριο ελπίζω ξέρω ότι ε, έχει φωνάξει κόσμο τους στρατηγούς, τους στρατιωτικούς ε, αυτό είναι για, ένα θέμα για το, για αυτό είναι ένα θέμα μόνο υπάρχουν και άλλα, και άλλα πολλά όσον αφορά την άμυνα γι' αυτό και το θέμα των σχέσεων με τη ΣΥΠΑ όσον αφορά την άμυνα θα πρέπει να μείνει ανοιχτό τόσο να μπορούμε να επανέλθουμε μια που ο κ. Ζωπάμα και η κυβέρνησή του σιγά σιγά θα διαμορφώσουν προτάσεις αλλά και πολιτικές. Εμείς ευχαριστούμε. Άλλοι δημιουργείς το λόγο. Εγώ πρόεδρε για να συμπληρώσω αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος ο Τομπίας Φρίγκερ έχω να σας πω ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να είναι τέτοια που να μπορεί να έχει περιθώριο να είναι ρεαλιστική και να φτάσουμε στο σημείο 0 για τους εξοπλισμούς, δηλαδή στον αφοπλισμό. Ακόμα όμως έχουμε πολύ δρόμο, ούτως ώστε να θεωρήσουμε ότι με μια τέτοια έκθεση θα καταλήξουμε σε μια ρεαλιστική πολιτική η οποία να προσφέρει στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα αυτή τη δυνατότητα του να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε. Γιατί ξέρουμε ότι μεσούντος του προσυγχρού πολέμου. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα όσον αφορά το να πετύχει κανείς κάτι τέτοιο. Γιατί τώρα πού πάμε, πάμε ανάποδα, πάμε στον επανεξοπλισμό. Αγνοούν αυτά που λέει ο ΙΕ. Κοφεύουν σε διάφορα τα οποία ακούγονται από επώνυμους, ας πούμε και στο Μόναχο. Όλοι όσοι πήγαν εκεί πέρα, ενώ ελέγχθη ότι με το 1% από τα όπλα να δώσει κανένα για το θέμα τη πείνα, θα το λύσει το πρόβλημα τη πείνα. Παρακαλώ. Λάβετε το υπόψη αυτό. Μην έχουμε επανεξοπλισμό. Αύξηση λέει των πολεμικών δαπανών. Δεν θα το είχαμε αυτό εάν. Εάν το, το, το, το, το σύνολο ε, στρατοκρατών, ΝΑΤΟ κλπ. εάν κάτι κάνανε. Αν είχαν εξυπηρετήσει σε κάτι τουλάχιστον. Δηλαδή σε Μπεσλάν, Μαδρίτη, Νέα Υόρκη, Γάζα, αν κάτι είχαν κάνει και δεν είχαμε αυτά που είχαμε. Η στρατιωτική αποτροπή δεν έκανε τίποτα. Πώς να τον κανένα να υπερασπίζεται ακόμα τέτοια, τέτοια ζητήματα. Γιατί το 99 είχαν αυτή τη νέα σύνθεση πραγμάτων ΝΑΤΟ είπαν λοιπόν ότι θέλουν να έχουν απάντηση θετική στον, ε, στην τρομοκρατία, στην ε, λαθρομετανάστευση, στο οργανωμένο έγκλημα, ε, να προσφερθούν κάποιες εγγυήσεις. Πού είναι λοιπόν αυτά τα οποία απαιτεί ο αιώνας μας από την ανθρωπότητα. Δεν νομίζω ότι έγινε τίποτα. Είδαμε στη Γάζα Πού φτάνει η πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Όταν αποφάσισαν οι Ισραηλινοί να χτυπήσουν τους στόχους τους. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιες λύσεις. Δεν θέλουμε να έχουμε σύστημα ασφαλείας το οποίο είναι προσδεδεμένο στο Αμερικανικό άρμα. Να μην είμαστε ένας παθητικός ε, μάρτυρας των εξελισσομένων πραγμάτων θα πρέπει να έχουμε δική μας θέση αλλιώς είναι θλιβερή η πολιτική μας γιατί έτσι δεν πάμε για δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου η Υπουργή Ασφάλειας θα πρέπει να χαρακτεί από εμάς τους ίδιους έτσι να βοηθήσουμε να γίνει εφοπλισμός έτσι να βοηθήσουμε να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο και βέβαια θα πρέπει να βοηθήσουμε τόσο ώστε ασφάλεια να σημαίνει αποστρατικοποίηση. Άρα λοιπόν, αλλά εμεί θα ψηφίσουμε αρνητικά και σε αυτή την έκθεση και στην έκθεση που ακολουθεί σε σχέση με ΝΑΤΟ και ΕΕ. Ο κύριος Λαντσμπέργκης, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ διαφωνώ κάθετα με την ε, προφορική ε, τροπολογία που κατέθεσε ο κύριος Κούνε Όπως και με πολλές άλλες τροπολογίες ε, για τις ε, χώρες της Βαλτικής. Γιατί όλα αυτά βασίζονται ε, σε ιδέες που μοιάζει να τις έχει παρουσιάσει ο κύριος Λαφοντέν. Αν κάποιος σου επιτεθεί και εσύ ενδιαφέρεσαι να αμυνθείς, εσύ είσαι ένοχος. Πρόσφατα η Γεωργία παρουσιάζεται ως ε, απόλυτα ένοχη για το ότι έχασε κατεχόμενα εδάφη και αγνοούμενους πολίτες. Και η Γεωργία σήμερα ε, μοιάζει να μένει απ' έξω από ένα νέο μέσο άμυνας. Φαίνεται αυτή είναι η εντολή του Κρεμλίνου για όλες τις χώρες που θα μπορούσαν να προμηθεύσουν όπλα στην Γεωργία. Οι χώρες της ε, Βαλτικής ε, όμως ε, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με την αλληλεγγύη που επιδεικνύουν. Μετά από μία κυβερνοεπίθεση και ραδινεργό επίθεση στο Λονδίνο την δολοφονία των Βρετανών πολιτών και τέλος τον πόλεμο σε αυτό που η Ρωσία αποκαλεί μετασοβιετικό χώρο, το ΝΑΤΟ επιτέλους ξύπνησε και τώρα σκέφτεται ε, το τι πρέπει να κάνει ε, στην περίπτωση άμυνας των χωρών της Βαλτικής. Αν τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαφωνεί, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σαφήνεια, απλά θα ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά μόνο στο ΝΑΤΟ. Ο κύριος Σαλαφράνκα, παρακαλώ, αν έχετε τη δυνατότητα να είστε σύντομος, γιατί έχουμε άλλη μια έκθεση να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο. Θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να θέσουμε από στρατηγική άποψη, να τοποθήσουμε στρατηγικά αυτή την έκθεση. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να κάνουμε σύγχυση μεταξύ του συγκυριακού και του θεμελιώδους. Ελέγχθη ότι η έκθεση δεν αναφέρεται στην ασφάλεια των πολιτών. Νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως εσφαλμένο. Δείτε στην πρώτη παράγραφο λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια κέπα η οποία να προστατεύει την ασφάλεια των πολιτών της και να προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα λέγεται ότι το πλαίσιο στο πρίσμα των απειλών θα πρέπει να αναθεωρηθεί σε συνάρτηση με αυτές τις απειλές τόσο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της ε, Διατλαντικής Συμμαχίας. Και είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ε, παγιώσει τις, ε, το δυναμικό άμυνας, παγιοποίηση, δεν το έχει συγκροτήσει και η πραγματικότητα είναι ότι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 27 μέλη, στήριξαν αυτούς τους στόχους στο πλαίσιο της, στρατηγικής, της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας. Αυτή η έκθεση νομίζω συμπεριλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία, κύριε Πρόεδρε. Ε, σηματοδοτεί τα ενδιαφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκαθιδρεί νέες σχέσεις με τη Ρωσία και συγκροτεί κάποιες ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε μια μορφή που επιθυμούν οι πολίτες. Κύριε Πρόεδρε, αν υπάρχουν πολιτικά θέματα θα πρέπει να τα, το αναγνωρίσουμε, όπως το θέμα της αντιπυρευλικής ασπίδας υπό το πρίσμα της πανεγικής ομιλίας του Ομπάμα. Νομίζω ότι μπορούμε να κρίνουμε κάποια πράγματα στην έκθεση, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά ξεκάθαρη. Και αύριο, η αυρινή μέρα θα κρίνει τα δύο ή τρία σημεία επί των οποίων υπάρχει διχογνωμία εδώ σε σχέση με την έκθεση αυτή. Και νομίζω ότι η Επιτροπή θα αποφασίσει με φρόνηση. Αλλά νομίζω ότι όταν ζητούμε κοινοβουλευτικό έλεγχο της ΚΕΠΑ το Κοινοβούλιο δεν υποστηρίζει μια έκθεση η οποία βάζει στο επίκεντρο την κοινοβουλευτική διάσταση και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο είναι λάθος. Γιατί ε, νομίζω ότι αυτό το απαιτούν οι πολίτες. Αλλιώς πραγματικά ε, προκαλούμε σύγχυση, συγχαίουμε το τυχαίο, το συγκυριακό με το θεμελιώδες όπως σας είπα στην αρχή. Ο κύριος Φων Βογκάου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση Νομίζω ότι με τις 200 ε, τροπολογίες που κατατέθηκαν φτάσαμε τώρα σε τρία μόνο σημεία που παραμένουν επίμαχα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω στον αλφο κύριο Κούνε ε, θα μου άρεσε πάρα πολύ να ε, καταργηθούν, να απαλληφθούν οι επαναλήψεις αλλά αυτό δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τα αποφύγουμε. Τα έχουμε πει στο παρελθόν, τα λέμε και τώρα γι' αυτό όλα αυτά εκφράστηκαν μέσα από τις τροπολογίες. Αυτά που είπε σχετικά με τον κυβερνοπόλεμο, cyber Ευχαριστώ Ευχαρίστως ε, να βρούμε κάποιον άλλο όρο. Cyber warfare σίγουρα να μην είναι ο καλύτερος όρος. Cyber attacks ε, αν θέλετε, είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε και με τον συνάδελφο κύριο Δημητρακόπουλο, ο οποίος ε, τοποθετήθηκε πάνω σε αυτό το θέμα. Νομίζω όμως ότι τελικά θα μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση. Κατόπιν υπάρχει το θέμα των χωρών της Βαλτικής. Υπάρχουν δύο θέματα εδώ. Η πρόταση του κύριου Βόγκαου λέει ότι πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός και ο κύριος Κούνε λέει τα ίδια. Όμως ε, τόσο συγκαλυμμένα του κύριου Κούνε που εγώ ως ε, απλός ε, πολίτης δεν θα μπορούσα να τα καταλάβω. Εγώ λοιπόν είμαι υπέρ της ξεκάθαρης συζήτησης και θεωρώ ότι αν τελικά αυτή η ξεκάθαρη συζήτηση δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία τότε έχουμε ως ε, καβάντζα την ε, πρόταση του κυρίου Κούνε. Τώρα, όσον αφορά ε, τον όρο missile defense, εδώ υπάρχουν διάφορες απόψεις. Άκουσα σήμερα τον κύριο Σβάτσενμπεργκ... και δεν είναι σίγουρο το τι θα κάνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Το μόνο που λέει η εκθεσή μου είναι ότι αν τελικά πράγματι αναγερθεί αυτή η αντιπυραυλική ασπίδα, τότε θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να ληφθούν υπόψη τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Αυτά λέει κατ' ουσίαν το άρθρο, με συγχωρείτε, το οποίο προτείνω. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νταφ για τις παρατηρήσεις του. Νομίζω ότι η Γαλλική Προεδρία ε, βεβαίως και ε, σφραγίστηκε από τον πόλεμο της Γεωργίας που τον χειρίστηκε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν όμω και άλλα θέματα που προχώρησαν. Η έρευνα, η άμυνα ε, στο Τσάντ παρά τις δυσκολίες ε, κατορθώσαμε να επιτύχουμε ένα αποτέλεσμα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να τα κρίνουμε όλα έτσι κάπως αντικειμενικά. Όσον αφορά την έννοια human security Ήδη κατά την τελευταία έκθεση διαφωνήσαμε. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτός ο όρος human security είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ακόμα ακριβώς όπως και ο όρος ευθύνη για προστασία, responsibility to protect. Εγώ όμως διαφωνώ το να αιτιολογεί κανείς ε, τις στρατιωτικές επιθέσεις με αυτή την πρόφαση. Υποτίθεται responsibility to protect. Και περιέργως πώς, εδώ συμφωνώ με τον συνάδελφο κύριο Φλούγκε. Νομίζω λοιπόν ότι πράγματι χρειαζόμαστε εδώ μία συζήτηση σε βάθος. Αυτά ε, για την ε, Γεωργία. Κατά τα άλλα, στην αρχική διατύπωση της εκθεσής μου η Γεωργία δεν αναφέρεται καθόλου. Λάθος βέβαια αυτό. Και τώρα πλέον προσπαθώ με μια προφορική τροπολογία να βρω μια διατύπωση η οποία αν θέλετε δεν είναι τόσο προχωρημένη όπως αυτή που έχει κατατεθεί και ε, αποδίδει κάποιες ευθύνες. Αν όμως μου δώσετε χρόνο μέχρι αύριο το πρωί θα προσπαθήσω και θα χαιρόμουν πάρα πολύ αύριο το πρωί αν είναι δυνατόν να συζητήσω και με τους εσκιώδεις εισηγητές για τα ανοιχτά, τα εκρεμή θέματα έτσι ώστε ή δυνατόν να καταλήξουμε σε μια κοινή πρόταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Η ψηφοφορία είναι αύριο και πάμε τώρα στην τρίτη έκθεση που και αυτή είναι ε, στενά συνδεμένη με τα προηγούμενα. Πρόκειται ε, για το ρόλο του ΝΑΤΟ στην αρχιτεκτονική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγητής είναι ο κύριος Βατάνεν. Πόση ώρα έχουμε, Πρόεδρε? Συνολικά ένα πεντάλεπτο. Δέκα ή δώδεκα λέει ο Πρόεδρος. Αλλά αν προτιμάτε να το κάνουμε αύριο το πρωί. Ίσως είναι πιο λογικό, λέει ο κύριος Βατάνεν, για να είμαστε δίκοι. Όχι γιατί το λέω εγώ. Το αξίζει αυτή η έκθεση. Περισσότερο χρόνο. Έχετε δίκιο, λέει ο Πρόεδρος, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σωστά τα λέτε. Επομένως, αύριο αρχίζουμε 9 ώρα με την έκθεση Βατάνεν. όλοι τώρα στην τηλεόραση να δούμε τον Ομπάμα.